start, we start, huh? Yeah. Good afternoon. I am opening the session, even waiting for those who are not yet here. Um, I have to ask for... Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η κυρία Βεργιέ και ο κύριος Ταβάρες έχουν προτείνει την ε, δυνατότητα για μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα της απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να κλείσει πρόθεσμα και χωρίς προειδοποίηση την ελληνική δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία. Επίσης υπάρχει μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό 2014 που θα είναι πιο σύντομη από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Το θέμα αυτό για την Ελλάδα λοιπόν μπορούμε να το δούμε αύριο το πρωί και έτσι μπορούμε να δούμε και το επόμενο μας θέμα που αφορά και πάλι τα τηλεοπτικά, ραδιοτηλεοπτικά. Έχετε καμία αντίρρηση, όχι. Κύριος Μέντες Δεβάλε θα πρέπει αύριο στις 10 να πάει στην ΑΦΕΤ για μια ψηφοφορία σε έκθεση της αρμοδιότητάς του και γι' αυτό θα πρότεινα να δούμε λίγο νωρίτερα τη δική του έκθεση για την ενέργεια των νέων στην ψηφοφορία. Να έρθει πρώτη δηλαδή, αν δεν έχετε αντίρρηση αύριο το πρωί. Δεν έχετε αντίρρηση. Καλώ. Εγκρίνουμε λοιπόν το σχέδιο ημερησίας διατάξεων. Διερμηνία υπάρχει εκτός από τα σλοβενικά, τα σλοβακικά και τα πορτογαλικά λέει η ομιλήτρια, όλες οι άλλες γλώσσες ε, εκπροσωπούνται. Δεν έχει αύριο σλοβακικά. Τώρα έχει σλοβακικά, δεν έχει σλοβενικά και πορτογαλικά. Και δεν υπάρχουν επίσης σουηδικά, φιλανδικά και άλλες, ε, σουηδικά, ουγγρικά και άλλες γλώσσες. Ούτε πορτογαλικά υπάρχουν. Λοιπόν, δεν έχουμε διερμηνία για τα πορτογαλικά. Μπορείτε να ακούτε τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ισπανικά. Μπορεί να μιλήσει Πορτογαλικά όχι, αγγλικά. Καλώς και στο συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος, αλλά... Αν δούμε και πώς είναι οι παριστάμενοι και πώς είναι συνήθως οι παριστάμενοι, τους ε, διερμηνείς τους φέρνουμε για το τίποτα. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα για είναι εκπαίδευση και τον αθλητισμό. έχουμε το δότηση από το κεφάλαιο 4, από το κεφάλαιο το σχετικό με τις εφαρμοστικές πράξεις. Έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε πριν από το καλοκαίρι σε μια συμφωνία. Θα συνεχίσω να σας ενημερώνω και ίσως μέσα στην εβδομάδα να δώσω και πιο λεπτομερείς απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες τώρα. Το θέμα των εγγύσεων δανείων και των κατεξουδόξεων συμπράξεων κάναμε ό,τι μπορέσαμε να τα συζητήσουμε, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει αποτελέσματα, πάντως αισιόδοξη παραμένω. Αυτά είχα να σας πω. Ερωτήσεις δεν έχετε. Σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη. Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης. κατερνά Νεβεντάλοβα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μου επιτρέπετε να μιλήσω σλοβακικά. Σήμερα καταθέτουμε την έκθεση για τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης η οποία στηρίζεται σε προτάσεις που απορρέουν από μια ευρύτερη συζήτηση που είχα προσπαθήσει να ε, αναπτύξω με εκπροσώπους από οργανώσεις και τα 25 μπλεκόμενους φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στην, ε, στις απαρχές αυτής της διαδικασίας είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις προτάσεις τους και έτσι καταλήγουμε στο, ε, στην έκθεση αυτή και τις προτάσεις μου που συνέταξα σε συνεργασία με τη Γραμματεία και άλλους φορείς. Αν αναφερόμαστε στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2012, ένα σχεδιασμό λοιπόν της εκπαίδευσης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων με αποτελέσματα και σε οικονομικούς όρους, με τρία έγγραφα. Εφτά έγγραφα εργασίας σε διάφορες κατηγορίες και θέματα. Ε, τα έχουμε χωρίσει έτσι γιατί είναι περιορισμένη η έκταση των εγγράφων εργασία αναγκαστικά λοιπόν. Και ξέρετε ότι στο θέμα της εκπαίδευσης υπάρχουν πολλά ζητήματα. Προσπάθησα να επικεντρωθώ πρώτον στην ανεργία των νέων και την στήριξη της απασχολησιμότητας χάρη στην εκπαίδευση. Γιατί ξέρετε είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα της ενεργείας. Έχει φτάσει στο 23% το Μάρτιο με τα στοιχεία που έχουμε. Άρα ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί να επανασχεδιαστεί η εκπαίδευση ώστε όταν τελειώνει ο νέος στις σπουδές του να μπορεί να βρίσκει μια θέση εργασίας και οι δεξιότητες οι οποίες αποκτά να έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Ε, θέλησα να επισημάνω ιδιαίτερα το διαδικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης που αξιοποιείται ο σύστημα σε αρκετές χώρες με πολύ καλά αποτελέσματα όπως η Γερμανία και η Αυστρία, με πολύ καλά αποτελέσματα, θεωρητική δηλαδή και πρακτική κατάρτιση και εκεί έχουμε τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων και επίσης εξυγχρονισμό του πεδίου δεξιοτήτων, γιατί είναι αρκετά πεπαλαιωμένα ακόμη, πρέπει κανείς να μάθει και να μαθαίνει και να μελετάει, πώς θα μαθαίνει και θα μελετάει και βέβαια να βελτιώσουμε, θα πρέπει να βελτιώσουμε και τις γλωσσικές δεξιότητες και άλλες. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε επίσης την απόκληση μεταξύ των οραμάτων των νέων ως προς τις σπουδέ τους ή την μετέπειτα ζωή τους και της πραγματικότητας με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι στην αγορά εργασίας και τις περιορισμένες ευκαιρίες που τους προσφέρονται. Να ζητούμε λοιπόν μία μέση οδό, ώστε να βοηθήσουμε τους νέους να διαμορφώνουν ρεαλιστικά οράματα. Και βεβαίως θα πρέπει να μπορούμε να τους καθοδηγήσουμε σωστά. Μια άλλη στόχευση είναι οι εταιρικέ σχέσεις με βελτίωση των συνεργασιών στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργασίες σε διάφορες χώρες. με την ε, συμμετοχή παραδείγματι του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος επιτρέπει την επαγγελματική πρακτική κατάρτιση στους νέους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και νέες σύγχρονες δεξιότητες, έτσι ώστε να βοηθούνται και οι ίδιοι αλλά και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προσανατολίσουν πως ότι θα πρέπει να διδάξουν στους νέους. Ένα άλλο ζήτημα είναι η συνεργασία με τον ε, τομέα των μη κερδοσκοπικών, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, εν ολίγης, όπου μπορούν να προσφέρουν ε, δυνατότητες απασχόλησης και κατάρτισης για τους νέους στον τετογενή τομέα και την απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων που θα μπορέσουν στη συνέχεια στον επαγγελματικό τους βίο να χρησιμοποιήσουν οι νέοι. Αυτού του είδους την εμπειρία λοιπόν, την επαγγελματική εμπειρία, μπορούμε να την προβάλλουμε και να την αξιοποιήσουμε περισσότερο. Χρειάζεται να υπάρξει ικανοποιητική αναγνώριση αυτής της εμπειρίας λοιπόν. Επίσης η ε, εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις έννοιες του ενεργού πολίτη, της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά ε, και έτσι θέλουμε να προβάλλουμε και τις ιδέες της εταιρική κοινωνικής ευθύνης για τις ε, επιχειρήσεις οι οποίες αν θέλουν να έχουν προσωπικό που θα είναι ικανό να εργαστεί στο μέλλον θα πρέπει και αυτές τις εταιρικές σχέσεις να υποστηρίζουν ώστε να ε, προσανατολίζεται εγκαίρως η εκπαίδευση στις ε, ανάγκες των επιχειρήσεων και να μην βρισκόμαστε με πολλές θέσεις εργασίας κενές για τις οποίες όμως δεν υπάρχουν κατάλληλοι υποψήφοι. Ένας άλλος τομέας είναι αυτός της διαβίου μάθησης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, όπου προσπαθώ να δώσω την έμφαση. Γιατί και η εκπαίδευση είναι βέβαια πολύ σημαντική, αλλά βλέπουμε ότι η επαγγελματική κατάρτιση παίρνει όλο και μεγαλύτερη σημασία. στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού δε, τους, τα άτομα με αναπηρίε, του ηλικιωμένους, τι γυναίκες, θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε να ενισχυθεί η δική τους συμμετοχή. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν και τα αναφέρουμε στις εκθέσεις μας. Και πρέπει να επικεντρωθούμε στο είδος της εκδίκευσης και των δεξιότητων που θέλουμε για το μέλλον, ώστε να διαμορφώσουμε το πεδίο το μαθησιακό που θα προσφέρει η εκπαίδευση. Με συγκεκριμένα βήματα, ώστε και ο ενδιαφερόμενος να βλέπει στην πράξη τι θέλουμε να του προσφέρουμε, τι προσπαθούμε να του προσφέρουμε, ώστε να μένουν τα πράγματα αυτά στη θεωρία, αλλά στην πράξη. γιατί υπάρχουν πολλά προγράμματα όπως ε, το σύστημα εγγύησεων για την νεολαία και δυνατότητες που προσφέρονται, τις οποίες θα πρέπει να συζητήσουμε, πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά και τις προκλήσεις πριν αυτές επιδεινωθούν. Πρέπει λοιπόν να στρέψουμε το κλέμα στο μέλλον, ταυτόχρονα όμως μην παραβλέποντας και τα προβλήματα της, ε, του παρόντος. Αυτά. Ε, περιμένω να ακούσω τι παρατηρήσεις σα, να δω τι τροπολογίες σας, Ελπίζω ότι δεν θα είναι υπερβολικά επικριτικές και θα με υποστηρίξετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σάντσες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήμουν εκπαιδευτικό και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή μας μάλλον και η έκθεση της Κατερίνα βάζουν την εκπαίδευση εκεί που της αξίζει. Θέλω να τη συγχαρώ λοιπόν για την εργασία της. Απαιτείται χρόνος βέβαια και πολύ παιδαγωγική προσπάθεια που μας λείπει έτσι ώστε η εκπαίδευση να σταθεί στο επίπεδο των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας που κάναμε εξ αρχής αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε δεσμούς ανάμεσα στην εκπαίδευση και τον χώρο της εργασίας. Κόσμους οι οποίοι είναι μερικές φορές στεγανοί και θα πρέπει οι ικανότητες τους οποίες θα δίνει το σχολείο να ανταποκρίνονται στις κοινωνικο-οικονομικές απαιτήσεις. Δεν υπάρχουν λύσεις σταύματα. Η δυσκολία είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να επιβαρύνουμε το κόστος της και να προσαρμοστούν οι ικανότητες που προσφέρει όπως είπαμε στις απαιτήσεις και όχι μόνο στην αγορά, στην αγορά εργασίας αλλά αυτό είναι απαραίτητο για όλους όσους χρειάζονται κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής ένα αναπροσανατολισμό της προσπάθειάς τους της εργασιακής. Η ανεργία θίγει τους νέους αλλά και από την άλλη υπάρχουν πολλές θέσεις που δεν μπορεί να καλυφθούν. Ε, υπάρχει δηλαδή μια αναντιστοιχία ανάμεσα τα αυτά που δίνει η εκπαίδευση και σε αυτά που χρειάζεται η αγορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει, να διευκολύνουμε δηλαδή την πρόσβαση στην αγορά. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη σε αυτά που έχουν στο νου τους ε, οι φοιτητές για τη δουλειά που θέλουν και στις ανάγκες της αγοράς ε, και στις φιλοδοξίες που είναι αναντίστοιχες με τις ικανότητες. Λοιπόν, χρειάζεται το θέμα της απασχολησιμότητας και του επαγγελματικού προσανατολισμού να μας απασχολήσει και χρειάζονται επίσης νέες εταιρικές συμφωνίες, σχέσεις, χρηματοδοτήσεις Ξέρουμε ότι και σε επίπεδο επαγγελματικών χώρων και σε επίπεδο εναλλακτικών μορφών επασχόλησης έχουμε πολλά να μάθουμε. Σε κάποιες χώρες έχουν υπάρξει βήματα προόδου όπως στη Γερμανία, στη δική μου χώρα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Εγώ ήμουνα καθηγήτρια Αγγλικής και γνωρίζω τη σημασία που έχουν οι γλωσσικές γνώσεις που πρέπει να επιτρέψουν στους Ευρωπαίους πολίτες να ωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα της κινητικότητας που θέλει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε λοιπόν την γλωσσική ικανότητα των νέων. Κάθε Ευρωπαίος πολίτης έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση και αν θέλουμε το δικαίωμα αυτό να γίνει πραγματικότητα, αυτό είναι ο στόχος μας, θα πρέπει να επενδύσουμε στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Η πρόεδρος αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό. Ο Λίνκολν είχε πει το κόστος της εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλό. Για κοιτάξτε όμως και το κόστος της άγνοιας Λοιπόν, πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την προσπάθεια αυτή στο ύψος των φιλοδοξιών μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την προετοιμασία αυτής της ε, έκθεσης που την θεωρώ εξαιρετικά σημαντική για το μέλλον των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη. Νομίζω ότι θέτει τα σημαντικότερα ε, θέματα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Ωστόσο, εγώ θέλω να ε, εστιάσω σε ορισμένε παρατηρήσεις που τους θεωρώ πολύ σημαντικέ. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να είμαστε πραγματιστές, πολύ ρεαλιστικοί στην προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε αυτή την εποχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και ενώ ρεαλιστική όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στα εκπαιδευτικά συστήματα. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στα δημόσια οικονομικά των κρατών και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εφάνταστους τρόπους και καινοτόμους τρόπους για να βρούμε τις τρόπους χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Πρέπει να γίνει αυτή η χρηματοδότηση και πιο αποτελεσματική. Οι συνεργασίες μεταξύ του επιχειρηματικού τομέα και της εκπαίδευσης φαίνεται να είναι μια λύση. Ανοίγει η εκπαίδευση του εκπαιδευτικό σύστημα και συνδέεται με την επιχειρηματικότητα και αυτό το θεωρώ επίσης σημαντικό. Να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό επίσης σημαίνει να δώσουμε στη νέα γενιά τις δεξιότητες και τις γνώσεις που πραγματικά χρειάζονται και θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους ζωή. Χρειάζεται να μειωθούν δραματικά οι απλές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Γιατί, Γιατί σήμερα αυτές τις γνώσεις μπορεί κανείς να τις βρει με ένα απλό κλικ στο ίντερνετ. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στις βασικές δεξιότητες, χωρίς κανείς να έχει ένα ε, επαρκές επίπεδο αλφαβητισμού και γνώσης ε, ε, αριθμητικής ή γνώσης πληροφορικής, είναι αδύνατο να προχωρήσει την εκπαίδευσή του. Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Επιτροπής, ακόμα σήμερα πολλοί Ευρωπαίοι νέοι δεν έχουν τις βασικές γνώσεις ανάγνωσης γραφής και μαθηματικών, ενώ άλλοι δεν έχουν τις βασικές γνώσεις πληροφορικής. Υπάρχουν επίση κάποιε άλλε εγκάρσει, πιο γενικέ δεξιότητες που χρειάζεται κανείς, όπως την δυνατότητα επίλυση προβλημάτων, την κριτική σκέψη, που χωρίς αυτές κανείς ε, νέος δεν θα μπορέσει να προσαρμοστεί στην ταχύτητα με την οποία υπέρχονται διαλλαγέ στην κοινωνία σήμερα. Ο κόσμος αλλάζει. Μπορούμε να συγκρίνουμε και να δούμε στην Ασία το εκπαιδευτικό σύστημα να παρέχει ακριβώς αυτές τις δραστηριότητες που εμείς χρειαζόμαστε στους νέους. Ενώ η Ευρώπη αντιδρά πολύ αργά και χάνει ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την Ασία, με την Κίνα, με την Ιαπωνία, με τις Ηνωμένες Πολιτείε. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της χαμένης γενιάς που δημιουργείται εξαιτία της τεράστιας ανεργίας. Θεμελιώδης στόχος της Επιτροπής Επιδείας και Πολιτισμού δεν είναι να ασχολείται με τις τράπεζες ή με την κατάσταση της οικονομίας στην Ευρώπη, αλλά να αντιμετωπίζει την ανεργία. Μέσω του τομέα για τον οποίο είναι αρμόδια, δηλαδή την παιδεία. Πρέπει λοιπόν οι νέοι στην Ευρώπη να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δαξιότητες και γνώσεις για να μπορούν να επιβιώσουν σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ. Yeah, thanks. Ε, ε. Κυρία Τρούπελ, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την Κατερίνα πρώτα απ' όλα. Και όταν σε άκουσα να μιλάς, ο φίλο μου λίγο ανακάλυψα πάλι θέματα τα οποία είχαμε συζητήσει ως προς τις βασικές ε, δεξιότητες για την διαβίου μάθηση, την κάλυψη του χάσματος, ε, στην εκπαίδευση κτλ. Και γι' αυτό θέλω να πω ότι διερωτώ με, και αυτό το απευθύνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερο, γιατί ακολουθείτε τώρα αυτή την προεξέγγιση από, το, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα στη συζήτηση για βασικές δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες, μαθηματικές δεξιότητες, δεξιότητες μάθησης σε έναν κόσμο που αλλάζει όλο και πιο γρήγορα. Όλα αυτά λοιπόν τα αναλύουμε και τα αντιλαμβανόμαστε. Ε, το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε αυτό, το πρόβλημα είναι περισσότερο το πώς θα αντλήσουμε τα διδάγματα, πώς θα λύσουμε τα προβλήματα, αλλά το να λέμε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικέ είναι οι γλωσσικέ δεξιότητε, οι ψηφιακέ δεξιότητε και ότι βεβαίω πρέπει κανεί να γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, μου φαίνεται περιττό. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή να μου πει για άλλη μια φορά γιατί και πώ το κρίνετε τόσο κατεπήγον αυτό ω ανάγκη. Δεν μπορούσατε να έχετε μια πιο διαφορετική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση, την ε, διακυβέρνηση, την άντληση των πόρων. Διότι σε θέματα δεξιοτήτων νομίζω ότι έχουμε ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Και για σας κύριε Τσβέαρ και τη σύγκριση μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων της Κίνας που αναφέρατε σε σχέση με αυτά της Ευρώπης. Το σύστημα είναι ότι ο μαθητής πρέπει να μαθαίνει, να μαθαίνει, να μαθαίνει, να μαθαίνει διαρκώς αλλά εκεί που είναι πραγματικά η δημιουργικότητα και ο σεβασμός στη δημιουργικότητα ίσως θα πρέπει να πούμε ότι ακόμη δεν έχουν φτάσει στο απόγειο. Ίσως αυτό οφείλεται και στο σχεδιασμό του πολιτικού του συστήματος. Ας μην ε, υποτιμούμε λοιπόν και ας μην αποδίδουμε όλα μας τα προβλήματα στην ε, δημιουργικότητα, την απουσία αυτής από τα εκπαιδευτικά μας συστήματα, γιατί χάρη σε αυτή μπορεί κανείς να προσαρμοστεί σε έναν όλο και πιο ταχαίως αλλάζοντα κόσμο. Κύριε Τζίμερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι έχω ήδη διαμαρτυρηθεί στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, διότι έχω το δικαίωμα να εκφράζομαι στην μητρική μου γλώσσα, όπως κάθε βουλευτής. δεν είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζω εγώ ίδιες με αυτές των άλλων και ειδικά σε μια επιτροπή που μιλάει για πολυπολιτισμικότητα, πολιτιστική ταυτότητα, θέματα του πολιτισμού, είναι το ελάχιστο να έχω το δικαίωμα να μιλάω όπως ο καθένας στη γλώσσα μου. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους βουλευτές που είναι εδώ παρόντες, αλλά και τη διαφάνεια, διότι οποιοδήποτε θέλει να παρακολουθήσει τη ζήτηση αυτή, μέσω του webstream παραδείγματι, θα πρέπει να έχει το ίδιο δικαίωμα να την παρακολουθεί στη γλώσσα του. Έχω ήδη διαμαρτυρηθεί, θα το επαναλάβω. Θα να ενημερώσω την Επιτροπή σας για την έκθεση. Θα ήθελα να πω ότι σκοπεύουμε να διατυπώσω κάποιες τροπολογίες στην έκθεση κυρίως στις παραγράφους που αφορούν τα μέτρα λιτότητας και τις περικοπές στους προϋπολογισμούς των κρατών που αφορούν την εκπαίδευση. Στο σημείο Γ, στο σημείο 4, γιατί θα μιλούμε για δημόσιους προϋπολογισμούς των κρατών για την εκπαίδευση, θα πρέπει να κάνουμε λόγο και για το πρόβλημα που πολλές χώρες αντιμετωπίζουν λόγω της Τρόικα, το γεγονό ότι απολύονται δάσκαλοι από τη δημόσια εκπαίδευση. Σήμερα στην Πορτογαλία έχει κηρυχθεί γενική απεργία των ε, διδασκόντων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί αναμένεται η απόλυση 30.000 καθηγητών για το επόμενο έτος. Πολλοί άλλοι έχουν ήδη απολυθεί. Θα περικοπούν ακόμα 30.000 θέσεις εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τι είδους λοιπόν ποιοτική εκπαίδευση μπορούμε να έχουμε όταν κόβουμε 30.000 θέσεις καθηγητών. Όλη αυτή η ιδέα λοιπόν της εκπαίδευσης και της σχέσης μεταξύ καθηγητή και δασκάλου που πρέπει να είναι στενή έχει ανατραπεί Δηλαδή έχουμε τάξεις με πολλά παιδιά, πολλούς μαθητές, για ένα μόνο δάσκαλο, για ένα μόνο καθηγητή, πράγμα το οποίο υποβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης. Και η ιδέα του να συγκεντρώνονται περισσότεροι μαθητές σε ένα σχολείο, να κλείνουν δηλαδή σχολεία και να συγχωνεύονται, ήδη έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Όχι μόνο στις κοινωνικές, στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, αλλά και προβλήματα συγκρούσεων, γιατί είναι περισσότερο ο συγχρονισμό είναι πολύ πιο έντονο, ο συγχρονισμό πιο πολλών ανθρώπων μέσα στον ίδιο περιορισμένο χώρο. Το επίπεδο λοιπόν της ε, ε, εκπαίδευσης πέφτει και λόγω αυτού του φαινομένου και του φαινομένου της σχέσης μεταξύ μαθητού και καθηγητή και του κατά πόσον μπορεί ο καθηγητής βέβαια να παρακολουθεί τη δουλειά ενός μαθητή. Αυτό πρέπει να καταγραφεί. Με γνώμη όχι μόνο την ποιότητα στην εκπαίδευση, βεβαίως, αλλά και με γνώμονα το πρόβλημα της ενεργείας, διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι σωστό βέβαια να απολύονται τόσες δεκάδες χιλιάδες δάσκαλοι και στη συνέχεια να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την ανεργία. Είναι αντιφατικό αυτό. Αυτά λοιπόν θα καταθέσω τροπολογία. Κατά τα άλλα είναι εντάξει. Ευχαριστώ, Σαντιάγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Καταρίνα, γιατί θεωρώ ότι το προσχέδιο έκθεσης είναι πολύ ενδιαφέρον. Το έχουμε συζητήσει το ζήτημα πολλές φορές στην Επιτροπή μας. Ε, γνωρίζουμε τους αριθμούς, γνωρίζουμε ότι το ποσοστό της ανεργίας για τους νέους είναι 23% στην Ευρώπη συνολικά και στην Ισπανία συγκεκριμένα είναι διπλάσιο. Επομένω, να μην επαναλάβω αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε τώρα είναι να εστιάσουμε περισσότερο στην επαγγελματική κατάρτιση. Αυτή τη στιγμή έχουμε την αίσθηση ότι είναι ζήτημα δεύτερης κατηγορίας. Δεν είναι εξίσου σημαντικό, αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο σημαντικό από ότι Επίσης χρειάζεται η σύνδεση με το χώρο της βιομηχανίας και της, ε, των επιχειρήσεων. Το ανέφερε και η μαθηταρές. Επίσης ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στη γλωσσομάθεια. Τρέψτε μου να εκφράσω και μια πιο ε, προσωπική άποψη. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε, να βελτιώσουμε μάλλον το κύρος των καθηγητών στη δευτεροβάθμια επεκπαίδευση στα σχολεία γενικά, τους δασκάλους και τους καθηγητές, γιατί έχουν χάσει το κύρος τους και αυτό υπονομεύει ακόμα και τη δυνατότητά τους ε, να διαχειρίζονται την τάξη. Πρέπει να ε, ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα, πιστεύω, και ε, ίσως καταθέσω και μια τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ, Σαντιάκο. Ωραία, βέβαια η έκκληση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς νομίζεις μπορεί να εξασφαλίσει περισσότερο σεβασμό προς τους διδάσκοντες, προς τους καθηγητές. Μπορεί πάντα κανείς να εκφράζει την ε, ευχή, αλλά ήταν βέβαια στην εποχή μου δεδομένος σεβασμός. Όταν χρόνια αργότερα όμως πήγα να δω ποια είναι η κατάσταση στα σχολεία, διεπίστωσα ότι πολλά είχαν χαθεί. Και ούτε μπορούμε να τα ανακαλέσουμε, γιατί αν δεν έχει ο γονέας σεβασμό για το δάσκαλο, τότε δεν έχει ούτε και ο μαθητής. Άρα είναι ένα ζήτημα Διαφορετική γενιάς. Αλλά μπορούμε να το γράψουμε και αυτό, γιατί όχι. Η Επιτροπή τώρα. Η κυρία Μακκέλεν είναι εδώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω για τις θετικές αντιδράσεις γενικά του Κοινοβουλίου στην έκθεση αναφέρεστε στις δράσεις που και εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικές που θα καταστήσουν ιδιαίτερα την επαγγελματική κατάρτισή μας παγκοσμίου επίπεδου, να είναι ευέλικτη, να προσανατορίζεται σωστά, να μπορεί να αναγνωρίζει και να αποδίδει εκεί που χρειάζεται τις λεγόμενες εγκάρσιες γνώσεις και ικανότητες. Στόχος της προσπάθειάς μας ήταν να δώσουμε μια σωστή αντίληψη στις περιφέρειες, στις κυβερνήσεις κτλ. Γιατί οι επενδύσεις στην συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι χρήσιμες για το μέλλον και το οικονομικό και το κοινωνικό δεν θα πρέπει να μειώνονται οι πόροι στην επαγγελματική κατάρτιση γιατί χρειαζόμαστε το σύστημα, το εκπαιδευτικό για να πετύχουμε μια ε, ευημερία οικονομική και κοινωνική στο μέλλον στις χώρες μας. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας λοιπόν και εκφράζω την χαρά μου γιατί βλέπω ότι γενικά υπάρχουν θετικές απόψεις γύρω από την προσπάθειά μας. Αυτό το οποίο επανέρχεται σε όλους είναι η σημασία των εταιρικών σχέσεων. Μία τροπολογία η οποία μπορεί να γίνει δεκτή αφορά το 12. Λέει ότι η ανακοίνωση δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα εφαρμοστικά μέτρα και ακριβώς εδώ Νομίζω ότι το Erasmus Plus είναι ένα πρόγραμμα μέσα από το οποίο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στις στρατηγικές έτσι, συνεργασίες που θα φέρουν σε επαφή την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και όλους τους εμπλεκομένους στην κατάρτιση, την εκπαίδευση και την εκπαίδευση έτσι ώστε από κοινού το σύστημά μας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στην πραγματικότητα του χώρου εργασίας. Θα μπορούσα να σας ενημερώσω και για τις δράσεις που αυτή τη στιγμή έχουμε αναλάβει, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές για την επιχειρηματικότητα που θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο του 2013 καλύπτει θα έλεγα κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που έκαναν τα μέλη σας για την σύνδεση με τις επιχειρήσεις έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να κατανοούν και τις προσπάθειες τις εκπαιδευτικές. Έχουμε επίσης και τα λεγόμενα τους πίνακες αποτελεσμάτων στον τομέα των γλωσσικών. Η πολυγλωσσία είναι πολύ σημαντικό πράγμα και ελπίζω να κάνουμε σημαντικά βήματα προόδου κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Ε, οι εταιρικέ συμφωνίες και σχέσεις για τις επαγγελματικέ σπουδές. Νομίζω ότι και τη μαθητεία θα ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου και αυτό θα προωθήσει οι γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλά που ακούσαμε από εσά. Τα σχόλιά σας ήταν, που ακούσαμε από εσά και δεν ήταν καλά για τις προτάσεις μας. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας. Ευχαριστώ. Κύριε Τούπελ, θα ήθελα να ζητήσω ένα συγκεκριμένο θέμα στην Επιτροπή. Είπατε ότι οι επιπτώσεις της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της οικονομίας είναι πολύ σημαντική. Νομίζω ότι η αντίληψη αυτή ανήκει και στη στρατηγική 2020 αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εμείς θέλουμε να επενδύσουμε περισσότερα στην εκπαίδευση και τη διαμεθοριακή μορφή εκπαίδευσης και συνεργασίας. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για καλύτερη προσπάθεια, μεγαλύτερη προσπάθεια από τις επιχειρήσεις. Γιατί λοιπόν για μια ακόμη φορά λέμε τα ίδια και τα ίδια. Μήπως θα ήταν καλύτερο να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας κυρίως στην εφαρμογή αυτών που έχουμε αποφασίσει. Αυτά που μας είπατε δεν είναι καινούρια. Τα λέμε εδώ και αρκετά χρόνια και ε, η άποψή μου είναι ότι σε αυτά βασιζόμαστε στη στρατηγική του 2020. Το να επαναλαμβάνουμε λοιπόν τα πράγματα δεν κάνει τη ζωή των μαθητών και των επιχειρηματιών καλύτερη. Θέλετε να το σχολιάσετε αυτό. Βεβαίως λέει η Επιτροπή. Προφανώς και υπογραμμίζουμε ότι η ανακοίνωση αυτή φέρνει σε επαφή τις δράσεις τις οποίες πρέπει να αναλάβουν, οφείλουν να αναλάβουν οι χώρες μέλη έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση στην οποία βρισκόμαστε και στον τομέα της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να συνδυάσουμε τις δράσεις αυτές σε ένα επίπεδο, σε ένα έγγραφο, ένα πρόγραμμα δράσης έτσι ώστε τα συστήματα, τα εκπαιδευτικά να στηρίζουν την ανάπτυξη, την οικονομική και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Προφανώς και εμπνέουν και την στρατηγική 2020, αλλά παρόλα αυτά έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και έχουμε συγκεκριμένα εφαρμοστικά μέτρα που θα είναι χρήσιμα για τα κράτη-μέλη να αναλάβουν. Να μας πούν ακριβώς το τι θα κάνουν και πώς θα υποστηριχθούν σε αυτό που θα κάνουν από, την, από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να ότι ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ δεν έχω την ίδια πίστη και πεποίθηση. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Μέχρι τώρα, τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ισπανία και την ενεργεία των νέων εκεί. Υπάρχουν διμερείς σχέσεις δυνατότητες για βοήθεια. Ξέρω ότι η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, παραδείγματι, έχει συνεργασία για το θέμα της ενεργείας με την Ισπανία, με την Ισπανική, ώστε να προσφέρει βοήθεια. Αλλά έχουμε διαρθρωτικά ταμεία, έχουμε περιφερειακά ταμεία. Ε, υπάρχει περιπτώσει, ποια είναι η ορατή απόδειξη ότι αυτά τα ταμεία δίνουν, φέρουν αποτελέσματα και ότι χρησιμοποιούνται ακριβώς για αυτούς τους λόγους, φερειπίν στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση ενεργείας των νέων. Και ε, δεν ε, διαμαρτύρομαι για τα ωραία αυτά λόγια που βρήκε ο κύριος ε, Νταλόβα, αλλά, αλλά πρέπει να δούμε και πράξεις, όχι μόνο λόγια όσο έγιναν αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση, διότι δεν έχει πράξεις πραγματικά να επιδείξει, ε, ε, αφήνει τα θέματα στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να υλοποιήσουν προγράμματα, αλλά θα πρέπει να ε, επιμείνουμε περισσότερο στα ακριβώς τα μέτρα που χρειάζονται να είναι αυτά που θα αναλαμβάνονται, διότι αυτοί που ε, έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία έχουν πια γεράσει και δεν τους έχουμε δώσει βοήθεια. Πώς θα γίνει λοιπόν πρακτικά να βρούμε τον τρόπο να τους στηρίξουμε για να προχωρήσουν λίγο περισσότερο, για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την ανεργία των νέων. Δεν θα διαφωνήσω λοιπόν και θα υποστήριξω πλήρω, το είπε η Ήλγα. Ωραία τα λόγια, αλλά πια δεν έχω πίστη σε αυτά που λέγονται. Και ο κύριος Σιγκάλσκι έχει στήσει τον λόγο. Ας προχωρήσουμε λοιπόν με μεγάλη πεποίθηση σε αυτά. Πολύ σύντομα να πω. Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά για τον εκτευρισμό της Προέδρου. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε αποτελέσματα και ότι δεν αρκούν τα λόγια. Να απευθύνω μια προειδοποίηση, επιτρέψτε μου. τη δουλειά στους νέους δεν θα τη βρουν οι ε, κρατικοί αξιωματούχοι. Χρειάζεται η οικονομία να λειτουργεί. Χρειάζεται, με λίγα λόγια, να αλλάξει η δομή της οικονομίας, να λειτουργήσει η οικονομία προκειμένου να μειωθεί η ανεργία. Στη Γερμανία είναι 5% η ανεργία, ενώ σε άλλες χώρες είναι πάνω από το 20%. Γιατί, ε, αυτό δεν είναι επειδή η πολιτική στη Γερμανία είναι πάρα πολύ καλή. Ο λόγος είναι επειδή η οικονομία της Γερμανίας λειτουργεί. Άρα ίσως καλύτερα αντί τον εκνευρισμό μας να τον στρέψουμε αλλού. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που δημιουργούμε τα προβλήματα. Τώρα έχουμε προξενήσει, και ανοίξει μεγάλη συζήτηση, δεν θα μπορέσουμε να τη λύσουμε, αλλά θα δώσω το λόγο στην Κατέρνα για να ολοκληρώσουμε. Naozaj veľmi plodnú debatu. Ja som si poznámky a verím, že keď e, navrhnete poznámky... Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλου Ήταν πολύ επικοδομητική συζήτηση. Σημείωσα όλε τι παρατηρήσει και με την κατάθεση των τροπολογιών είμαι βέβαια ότι θα είμαστε θέση να τι αποδεχθώ με βάση τα όσα άκουσα σήμερα. Για το κείμενο η, προ... η παρατήρηση μου είναι ότι η πρόταση του Κοινοβουλίου καλή είναι. Είπατε, ας αν θέλει να μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε τις θέσεις της. πάρα πολύ καλό, ευχαριστούμε. Στο σημείο 12, το κείμενο της Επιτροπής συνεπάγεται ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Γι' αυτό η δική μας η παρατήρηση ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Καλό είναι να καταθέσετε και περαιτέρω προτάσεις για εταιρικές σχέσεις και το καθεξής, αλλά δεν ε, αφορά αυτό το κείμενο γιατί δεν έχουν υλοποιηθεί όλες αυτές οι εταιρικέ σχέσεις. Μακάρι λοιπόν να υλοποιηθεί κάτι πρακτικά και θα το δεχθούμε. Καλώς Κατέρνα, σε καταλάβαμε, λέει η Πρόεδρος. Το Σεπτέμβριο θα γίνει η ψηφοφορία. Προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών 27 ε, Ιουνίου, προσεχή εβδομάδα. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Τέσσερα ιστορική μνήμη στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μιγκάλσκι, Μάρικ Χένρικ. Δόκτωρ Μιγκάλσκι, έχετε τον λόγο από την Πολωνία. Ja rozpocznę ten, pierwszą wymianę poglądów. Ναι, Πρόεδρε, Θα ξεκινήσω με αυτό που ίσως είδατε και εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια έκθεση, όταν πηγαίνει κανείς προς την πλατεία του Λουξεμβούργου, βλέπει μια έκθεση η οποία οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ξεκινήσω από τις εικόνες που βλέπουμε. Θα ήθελα να αρχίσουν οι εικόνες να προβάλλονται Αυτές είναι οι πρώτες ε, εικόνες της παρουσίασης. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεννήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τη δραματική εμπειρία των δύο ολοκληρωτικών συστημάτων ή καλύτερα του πολέμου των δημοκρατιών εναντίον του ναζισμού. Πρόκειται για μια εμπειρία η οποία οδήγησε στο θαύμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δείτε τι έχει μεγάλη σημασία για μας. Το 46 σαν παράδειγμα, το 46 βλέπουμε την ελευθερία ενός τμήματος της Ευρώπης. Οι φωτογραφίες τις οποίες βλέπουμε εκτός του κτηρίου του Κοινοβουλίου το δείχνουν αυτό. Είμαι ευγνώμων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε την ιστορία της Ευρώπης σε καμιά δεκαριά εικόνες. Βλέπουμε την ουσία, από τη μία την ευημερία και την ειρήνη και από την άλλη βλέπουμε την ΕΚΑΧ Από την άλλη έχουμε λοιπόν την διέρεση της Ευρώπης. Βλέπουμε την επανάσταση στην Ουγγαρία το 1956. σε αυτή τη φάση αναπτύσσεται η Δυτική Ευρώπη, αλλά η Κεντρική Ευρώπη και η Ανατολική Ευρώπη παραμένουν κάτω από τον κομμουνιστικό ζυγό. Παράλληλα, όπως βλέπετε εδώ, πολύ συνοπτικά, ε, βλέπουμε ε, τα τελευταία 50 χρόνια της ε, ιστορίας της Ευρωπαϊκής. Δεν προετοίμασα εγώ αυτές τις εικόνες, δεν τις επέλεξα εγώ. Είναι ιδέα του ιδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπουμε εδώ τους Σλοβάκους, βλέπουμε την ευημερία στην Δύση, Βλέπουμε τον Βίλι Μπραντ, ο οποίος γονατίζει στη Βαρσοφία μπροστά στο μνημείο του γκέτο του εβραϊκού της πόλης. Βλέπουμε στην Ισπανία, τι συνέβη στην Πορτογαλία, η οποία Πορτογαλία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε την γερμανογαλλική ή γαλλογερμανική συμφιλίωση βλέπουμε την ενιαία Ευρώπη με την καταστροφή του ε, τείχους στο Βερολίνο. Μετά βλέπουμε κάποια συμβάντα, τα προβλήματα που είχαμε στις δεκαετίες του 70 και του 80 και φτάνουμε το 2004 που είναι μια πάρα πολύ σημαντική χρονολογία για την συμμετοχή των υπολείπων χωρών της Ευρώπης, της μετακομμουνιστικής Ευρώπης πλέον που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας αυτό είναι το πραγματικό τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. No i to są ostatnie dwa obrazy, które są tam na, na, tej, na tej antresoli przyznanie Unii Europejskiej. Και εδώ είναι οι τελευταίες εικόνες. Βλέπουμε το βραβείο Νόμπελ για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 12. Ja pokazałem to dlatego, żeby Państwu uświadomić, w którym kierunku, czy zaanonsować, w którym kierunku chciałbym pójść w... Γιατί σας τα δείχνω όλα αυτά. Μόνο και μόνο για να σας προσανατολίσω σχετικά με την παρουσίασή μου, να δείξω το διοικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που φτάνει θα έλεγα στην, κορύφωσή, στην κορύφωσή της το 2004. Να σας δείξω ότι πάρα πολλοί Ευρωπαίοι έχουν ξεκινήσει να ωφελούνται από την Ευρώπη μόνο στη δεκαετία του 80 ή του 90 μάλλον και ε, ήδη το 90 είναι για μας τμήμα της ιστορικής μνήμης, ενώ η ιστορική μνήμη των κατοίκων της Δυτικής Ευρώπης και της Ανατολικής Ευρώπης διαμορφώθηκαν με διαφορετικό τρόπο. Και οι δύο είναι σημαντικοί και οι δύο, ε, οι δύο περιοχές είναι σημαντικές. Ο ναζισμός ήταν μια πολύ σημαντική ιστορία για όλους μας, ενώ οι εμπειρίες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης ήταν λίγο λιγότερο καθολικές θα έλεγα, αλλά ανήκουν και αυτές στην ιστορική συλλογική μνήμη. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα στην έκθεσή μου να λάβουμε υπόψη μας τα θεμέλια της ευρωπαϊκής κοινότητας σήμερα, την συνοχή, την ανοχή, τον χριστιανισμό, την επιστήμη, το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Θα ήθελα όλα αυτά να αποκτήσουν ένα επιπλέον νόημα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε σωστά τις αξίες μας και να κατανοήσουμε ακριβώς σε τι πυλώνες έχει οικοδομηθεί ή ε, το παρόν, η ταυτότητά μας. Θα ήθελα λοιπόν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία με όλους όσους πάρουν μέρος στην ε, επεξεργασία της έκθεσης αυτής. Να μου πούνε με συγκεκριμένο τρόπο σαν παράδειγμα πώς θα υποστηρίξουμε όλες τις πρωτοβουλίες επιστημονικές ε, και πολιτικές που οδηγούν στην έρευνα της ιστορικής μνήμης να ζητήσω επίσης βοήθεια για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Μνήμης και Συνείδησης. Θα ήθελα να μην καταργηθούν μέσω των περικοπών α, τις υπηρεσίες στην Ευρώπη των πολιτών και θα ήθελα επίσης να υποστηρίξουμε και την πρωτοβουλία μας σε συγκεκριμένες ιστορικές πρωτοβουλίες που έχουν σαν στόχο την ίδια την ιστορική μνήμη. Πιστεύω επίσης ότι ό,τι σχετίζεται με τη συμφιλίωση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σαν παράδειγμα η γερμανική συμφιλίωση, η συμφιλίωση ανάμεσα στις δύο Γερμανίες, η συμφιλίωση ανάμεσα στην Πολωνία και τη Γερμανία. Ήταν πολύ σημαντικά θέματα και έδωσαν σχήμα και μορφή στην ιστορική πολωνική μνήμη. Πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να ανοίξουν τα αρχεία τους ε, και έτσι μόνο θα μπορέσουμε να αναλύσουμε την ιστορική μας μνήμη. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι η έκθεση αυτή να μην βασίζεται σε καινολογίες. Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους συνεισηγητές, σε όλους όσους συνεργαστούν μαζί μου, έτσι ώστε το έγγραφο αυτό να μην είναι ένα γενικόλογο έγγραφο που να βολεύει όλο τον κόσμο. Θα ήθελα με αφορμή το έγγραφο αυτό να μπορέσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεισφέρουμε στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στον τομέα της εκπαίδευσης και στον τομέα του πολιτισμού. Υπάρχουν κάποια έγγραφα στα οποία έχουμε ήδη αναφερθεί και γι' αυτό θα ήθελα η έκθεσή μου να είναι αληθής, να βασίζεται στην εμπειρία και να είναι μια καλή αφορμή για συζήτηση του κοινού μας παρελθόντος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μεράντα Τεβάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια. Έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να θέσουμε συγκεκριμένα θέματα και πράγματι η ιστορία με τις εικόνες είναι κάτι το οποίο μας ε, πάει πραγματικά πίσω. Σε μια ομιλία την οποία έκανε ο Χόρχε Σεμπρούν το 2010 για τα 60 χρόνια της απελευθέρωση των κρατουμένων του Μπούχενβαλτ, όπου ήταν ο ίδιος ο Ισπανός συγγραφέας ε, από το 1943 μέχρι το 1945, ο Σεμπρούν μας είπε ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσει να επηρεάσει υπαρξιακά και πολιτιστικά αν συμμεριστούμε και μοιράσουμε πραγματικά τις μνήμες μας και νομίζω ότι αυτή είναι και η γραμμή του κυρίου ε, Μιγκάλσκι. Δεν υπάρχει μία θα έλεγα ε, τέτοια ιστορία. Σε ένα πλαίσιο τώρα πολιτικής και οικονομικής κρίσης, στην οποία βιώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε ότι οι πανεπιστημιακοί διανοούμενοι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή οικονομικης κρισης την οποια βιωνουμε στην ευρωπαικη ενωση ξερετε οτι μνήμη. Αυτή η ιστορική μνήμη βέβαια συνεχίζει να διαμορφώνει όχι μόνο τις σημερινές διμερείς σχέσεις της Ευρωπαϊ... των μελών της Ένωσης, αλλά και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Το 2007 η καταστροφή ενός σοβιετικού μνημείου στο Ταλίν δημιούργησε μια κρίση ανάμεσα στην Εσθονία και τη Ρωσία. Αλλά μια διμερής κρίση ήταν αυτή, όχι μια κρίση ανάμεσα στην Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν ήταν κάτι που ανήκε στην κοινή ιστορική μνήμη της Ευρώπης, γιατί τότε θα υπήρχε μια συλλογική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταστροφή του συγκεκριμένου μνημείου. Πρέπει λοιπόν να καταλήξει κανείς σε μια πανευρωπαϊκή μορφή ιστορικής μνήμης. Πρέπει να συζητήσουμε και τα κοινωνικά και τα κοινά πολιτικά και, και τα κοινά κοινωνικά προβλήματα. Θα μπορέσουμε εφόσον τα παρουσιάσουμε με σωστό τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε μέσω αυτής της κοινή μνήμης. Θα πρέπει να πω ότι μέχρι τώρα ένας ορισμός της κοινής θα έλεγα μνήμης περιορίζεται θα έλεγα σε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Πέραν αυτών όμως που φυσικά δεν πρέπει να αγνοούμε τις λεπτομέρειες νομίζω ότι μια αφεντική ευρωπαϊκή ιστορία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πολιτικές απελάσεων, θα πρέπει να περιλαμβάνει την απικιακή ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την γενοκτονία των Αρμενίων και πολλά άλλα θέματα. Ο ανταγωνισμός και η ιεραρχία ανάμεσα στην μνήμη του Γκουλάγκ και τη μνήμη ε, της ΣΟΑ έχει οδηγήσει σε μια διέρεση θα έλεγα αυτή την κοινή ιστορική μνήμη. Ξέρετε ότι το θέμα της ΣΟΑ ε, θεωρείται, ε, έχει, είναι κάτι που έχει σχέση με την άρνηση της αναγνώρισης από πολλούς κάποιων εγκλημάτων από πλευράς της Σοβιετικής Ένωσης. Το βασικό εμπόδιο στη φάση αυτή για την κοινή μνήμη είναι η συμφιλίωση ανάμεσα σε μνήμες ανταγωνιστικές του Γκουλάγκ και του Ολοκαυτώματος. Εκεί βρίσκεται το θέμα. Ο Χόρχε λοιπόν, ο οποίος ήταν ε, παλαιά ε, όταν το κόμμα το κομμουνιστικό ήταν στην παρανομία, ήταν ο του και μετά έγινε ε, υπουργός πολιτισμού και είχε εκφράσει όμως την ελπίδα του, είχε πει ότι στην επόμενη επέτειο θα έλεγε κανείς ε, για τα 100 ίσως χρόνια του Μπούχενβαλ, το Γκουλάγκ θα έχει ενσωματωθεί και αυτό στην κοινή ευρωπαϊκή μνήμη. Η συλλογική ευρωπαϊκή μνήμη και τελειώνω εδώ παρουσιάζεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο όσο πολλές είναι και οι χώρες και δεν μπορεί να ενιοποιηθεί, να ενοποιηθεί συγγνώμη, μέσω των τελετών. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί από την επιθυμία μόνο των κοινοβουλίων αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να παρουσιάζουν τα εγκλήματα του παρελθόντος με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφύγουν την επανάληψή τους στο μέλλον. Η τάση που λέει ότι η λύθη είναι καλύτερη από τη μνήμη είναι κάτι που εφαρμόστηκε και στην μεταπικιακή Γαλλία και στη μεταφραγκική Ισπανία, πολλοί θα ήθελαν, και ίσως εν μέρη και στην μετακομμουνιστική Πολωνία. Αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να αρνηθούμε. Λέμε όχι στην αμνησία, όχι στη λύθη. Ο εκδημοκρατισμός των σε μετάβαση δημοκρατιών θα είναι ατελής εάν δεν μπορέσουν να δουν με κριτικό βλέμμα το παρελθόν τους έτσι ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη, αποκατάσταση και αναγνώριση. Η αδίποτε πρωτοβουλία για κοινή ιστορική μνήμη θα πρέπει να είναι υπεράνω κάθε προσπάθειας εκδίκησης. Μόνο αναγνώριση, μόνο δικαιοσύνη, μόνο ε, όχι ε, εκδίκηση, όχι πνεύμα εκδικητικό. Λοιπόν, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η δημιουργία μιας κοινή ευρωπαϊκής μνήμης πρέπει να είναι βασικό συστατικό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο κύριος Μιγκάλσκι το είπε ότι απαιτείται σαν προϋπόθεση η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των μεμονωμένων Ευρωπαίων πολιτών. Πέραν αυτό, η διαδικασία δημιουργίας της ιστορικής μνήμης είναι κάτι το πολιτιστικό και όχι αυστηρά παιδαγωγικό. Προαπαιτεί την αναγνώριση και ε, την προσπάθεια εμφύσισης κάποιων αρχών και αρετών. Δεν θα πρέπει εμείς απλά να επιβάλλουμε περισσότερες ώρες διδασκαλίας της ιστορίας, αλλά να μάθουν τα παιδιά την ιστορία και από άλλες δραστηριότητες εκτός σχολείου, από τη λογοτεχνία κτλ. Θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου μας, Πρόεδρε. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Μιγάλσκι και για την προσφορά συνεργασίας και για μια έκθεση η οποία έχω την αίσθηση ότι με τη δική σας ικανότητα κύριε Μιγκάλσκι μου θα είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ πολύ καλά κύριε Ντεβαλέβ. Έχετε πολύ καλά προετοιμαστεί για το θέμα αυτό. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Κοιτάξτε, είμαι σοβαρό άνθρωπο και έρχομαι προετοιμασμένο. Δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο αυτό που συνέβη. Πάντα είμαι σοβαρός. Όχι, μα δουλέψατε πάρα πολύ σοβαρά και μέχρι και θα ξεπερνούσατε τον κύριο Μιγκάλσκι σχεδόν. Χωρί μικρόφωνο κύριο Μιγκάλσκι η κυρία Σάντσο Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο και για την παρουσίαση του που ήταν πολύ συγκεκριμένη. Καταλαβαίνω πολύ καλά ποιες οι ανησυχίες του και την ε, επιδίωξή του να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες ενέργειες. Τώρα, από τη δικιά μου την πλευρά θα ήθελα να πω το εξή. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ιστορική μνήμη χωρίς να μιλάμε για την πολιτιστική κληρονομιά και αναφέρομαι στην ε, Ευρωπαϊκή ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μια πρωτοβουλία ε, κατά τη διάρκεια της οποίας οργανώνονται επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία με, που τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα το παρελθόν, το κοινό μας παρελθόν, την ιστορική μας μνήμη και την πολιτιστική μας ε, κληρονομιά. Φυσικά δεν μπορεί αυτό να γίνει μέσα από όλα τα, τα θέματα της εκπαίδευσης, αλλά πάντως η ε, πολιτιστική κληρονομιά αφορά όλους τους τομείς της ε, ε, εκπαίδευσης. Χρειάζεται οι μαθητές να εκτιμούν αυτήν την κληρονομιά. Και μοιράζομαι και εδώ και την προσωπική μου εμπειρία, το συναισθήματα και την συγκίνηση που προκαλεί στους μαθητές μια τέτοια επίσκεψη πόσο αυτό ε, βοηθά στο να εγγραφούν αυτές οι αξίες στο, στη συνείδηση των μαθητών. Το ζήτημα λοιπόν της πολιτικής κληρονομιάς είναι περίπλοκο γιατί αυτά τα μνημεία πολύ συχνά συνδέονται με παρελθούσες συγκρούσεις. Συγκρούσεις οι οποίες μπορεί να συνεχίζουν να δηλητριάζουν το παρόν. Γι' αυτό πιστεύω ότι η μνήμη και η πολιτιστική κληρονομιά μπορούν να συνδυαστούν για την ε, εκπαίδευση των πολιτών. Ο κύριος μας ζητά να βάλουμε στο κέντρο της συζήτησής μας την κοινή ε, ευρωπαϊκή ε, κουλτούρα και ε, υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης, ένα θέμα που γνωρίζετε ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καθώς επίσης και τη σημασία που έχει τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά από τη μικρότερη ηλικία μέχρι το πανεπιστήμιο η πολιτιστική κληρονομιά εξάλλου είναι κατά την απόψή μου ε, το καταλληλότερο μέσο για την προώθηση, προάσπιση της ιστορικής κοινή ευρωπαϊκής μνήμης. Πρέπει λοιπόν να αναφερθούμε σε ε, εκπαιδευτικές δραστηριότητες Κατά τη διάρκεια του 2014 θα διοργανωθούν διάφορες εκδηλώσεις ε, ιστορικής ε, μνήμης, ε, καθώς συμπληρώνονται και τα 60 χρόνια από τη λήξη ενός πολέμου σημαντικού για την ε, Ήπειρο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι Πρέπει να συγχαρώ μάλλον τον ε, κύριο Μιγκάλξη και μην πω ότι ζηλεύω και το γεγονό ότι ανέλαβε να συντάξει την έκθεση για αυτό το θέμα που είναι τόσο σημαντικό. Εμείς στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη ε, το, μας αγγίζει ε, αυτό το ζήτημα. Μόλις εχθές γιορτάσαμε τα γεγονότα στο Βερολίνο και στην Ουγγαρία. Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας ε, εκείνη την εποχή είχε εκτελεστεί στις 16 Ιουνίου. Και τα αναφέρω αυτό ως ένα παράδειγμα ενός συμβολικού γεγονότους που μπορεί να βοηθήσει την χτίσιμο της ιστορικής μνήμης. Αλλά βλέπουμε εδώ και τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της ιστορικής μνήμης και της ε, καθημερινής άσκησης πολιτικής. Πρόσφατα επισκέφτηκα την ε, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και διατυπιστώσαμε ότι ένα από τα προβλήματα στην ένταξη της ε, ΦΥΡΟΜ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι ιστορικές σχέσεις αυτής της χώρας με την Βουλγαρία και την Ελλάδα. Είναι ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Όπως βλέπετε λοιπόν πώς οι ιστορικοί πώς ιστορικά γεγονότα συνεχίζουν να επηρεάζουν ακόμα και σήμερα την άσκηση πολιτικής και πώς μπορεί να δημιουργήσουν ε, ε, προβλήματα ε, στην ευρωπαϊκή πολιτική. Το ίδιο ισχύει και για τις πληγές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πιστεύω λοιπόν στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής ιστορίας. Έχουμε παραδείγματα όπως η Σλοβακία, ε, η, η περίπτωση της Ουγγαρίας όπου η Ανάσταση του 1948 έχει ε, αποσιωπηθεί και η σύγκρουση μεταξύ Σλοβακίας και Ρουμανίας για ιστορικά γεγονότα. Συχνά. Και πολύ συχνά χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν μιλούμε από τη μια για τα τις αποτελέσματα του φασισμού και από την άλλη για τα αποτελέσματα του κομμουνισμού. Είναι δύσκολο λοιπόν να ε, ερμηνεύσει κανεί την ιστορία, αλλά ακριβώ γι' αυτό χρειάζεται η ευνοποίηση τη ευρωπαϊκή ιστορία, κατά την άποψή μου. Πολύ συχνά ακούγεται η άποψη ότι το σημαντικό είναι η οικονομία, ε, το εμπόριο και ότι η ιστορία έρχεται σε δεύτερο μοίρα. Διαφωνώ. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη επένδυση είναι η επένδυση στην ιστορία. Και ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ω οικοδόμημα ε, μπορεί να κοστίζει ακριβά, πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό να επενδύσει στην ιστορία, στην κοινή μα ιστορία, παρά στο πρόγραμμα Εράσμους, για παράδειγμα. Και όσον αφορά αυτήν την κοινή μα ιστορία, νομίζω ότι πρέπει μια και έξω να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και αυτές τις κρίσεις στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Εάν τα καταφέρουμε αυτό νομίζω ότι θα έχουμε τεράστια πολιτικά και άλλα πλεονεκτήματα. Ορισμένοι λένε ότι ε, στην Ευρώπη τίποτα δεν έχει αξία αλλά όλα έχουν την τιμή τους. Ε, εγώ από την πλευρά μου θα έλεγα ότι πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση και να μιλούμε για αξίες και όχι για την οικονομική διάσταση του κάθε πράγματος. αυτό το ζήτημα προφανώς εμπίπτει στο χαρτοφυλάκιο της Επιτροπής μας. Αυτά τα... Αυγούστου είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα ε, αναλυθεί μια πρωτοβουλία για την ιστορική ανάμνηση όλων των ε, θυμάτων δικτατοριών. Είναι ένα παράδειγμα τέτοιας επαιτίου. Με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ενοποίηση της υπήρους μας. Ευχαριστώ. Κύριε Τρίπελ, πρόεδρε, νομίζω θα πρέπει να αναφερθούμε σε κάτι που πάνε οι συνάδελφοι Μιγκάλσκι και Μερέντε Βάλε. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να, να αναγνωρίσουμε ότι υπήρξαν διαφορετικά ολοκληρωτικά συστήματα στην Ευρώπη. Τα επρόκειτο για εθνική κοσοσιαλιστικά, εθνικιστικά ε, ολοκληρωτικά συστήματα ή κομμουνιστικά ολοκληρωτικά συστήματα, χωρίς να θέλω να τα αξιολογήσω σε βαθμίδες. Ε, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας, δύσκολο κομμάτι της ιστορίας μας, όπως και η επικοιοκρατία. Και βεβαίως, από την άλλη πλευρά, υπάρχει η θετική ιστορία στην Ευρώπη, η διακήρυξη των ανθρωπινών δικαιωμάτων, που όμως έχουν παραβιαστεί επανειλημμένως και μην ξεχνάμε τη Σρεμπρένιτσα ως παράδειγμα. Ε, άρα λοιπόν έχουμε και τα χειρότερα, τα πιο φρικτά εγκλήματα, αλλά και τα ε, υψηλότερα ιδεώδη που έχουν περάσει από την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι εάν θέλουμε να μιλήσουμε για μια κοινή κουλτούρα μνήμης θα πρέπει να μιλάμε στον πληθυντικό γιατί είναι πολλές οι κουλτούρες μνήμης και ο κόσμος, ο πολίτης αισθάνεται πολλαπλά, ε, πολλαπλούς τραυματισμούς στην ιστορική του μνήμη για τον έναν είναι το ένα ιστορικό γεγονός διαφορετικό τραύμα από ότι τον άλλον. Άλλος γιατί ήταν πρόσφυγας ύστερα από πόλεμο εμφύλιο, άλλος γιατί ήταν θύμα της απεικιοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν η αυτοκριτική ή το ζήτημα της δυνατότητας σε ενδοσκόπηση και προβολή στην ιστορία της Ευρώπης και την ιστορία του κόσμου νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη σημασία στην υπόθεση αυτή. Νομίζω πάντως ότι όσο και να τονίσουμε το θέμα της μνήμης και της ιστορικής μνήμης, στις τωρινές συνθήκες των ρήξεων και των ε, αντιπαλωτήτων, των πολιτιστικών συγκρούσεων, γιατί μιλάμε ακόμη και τώρα για σύγκρουση πολιτιστική μεταξύ Βορρά και Νότου ενδεχομένως, ε, αγεφύρωτη ή για, το για τα όσα είπε ο κύριος Μελανσόν για τη Γερμανία και την ε, πολιτιστική απόσταση. Πράγματα τα οποία εμένα με τρομάζουν γιατί μας γυρνάνε πίσω σε ιστορία που η Ευρώπη θα έπρεπε να έχει αφήσει πίσω της και δείχνουν ότι δεν έχουμε μπορέσει να διδαχθούμε από τα σφάλματα του παρελθόντος και με όλες τις διαφορές που μεταξύ μας να εστιαστούμε στα ουσιώδες και σε αυτό που θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε το μέλλον μας καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω έκκληση να μιλήσουμε βεβαίως για τη μνήμη, για τη δουλειά αυτή της μνήμης και την κουλτούρα της μνήμης και την ενδοσκόπωση και να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τραυματισμοί και τραύματα που όμως έχουν οδηγήσει μπροστά, έχουν ε, συνυπάρξει μέσα σε αυτό το εγχείρημα της Ευρώπης. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι με την επεξεργασία αυτή τη ιστορική μνήμη μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η τωρινή κρίση που αντιμετωπίζουμε δεν πρέπει να μα ε, κάνει να χάσουμε από τα μάτια μα αυτό το, το θέμα, αυτή τη ε, διάσταση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ντελβάγε. Εξετίμησα δεόντως τα λεγόμενά του στα πλαίσια της ιστορικής εικόνας της Ευρώπης δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την απεικιοκρατία. Και απογοητεύτηκα γιατί στα πλαίσια της συζήτησης σχετικά με τη νομική βάση της Ευρώπης για τους πολίτες υπήρχε μια τροπολογία για την απεικιοκρατία πέραν του φασισμού και του σταλινισμού και δεν έγινε δεκτή. Πρόκειται για ένα τυφλό σημείο της ε, ευρωπαϊκής ιστορίας και ιδιαίτερα της Γαλλίας ελπίζω να επανενταχθεί στη συζήτηση. Έχει μεγάλη σημασία στα πλαίσια της ιστορικής αυτής εικόνας να εμείνουμε ε, στην ιστορική αυτή διάσταση της απεικιοκρατίας. Να πω εδώ ότι η δουλειά των ιστορικών είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κλειό. Είναι ένα δίκτυο ιστορικών που κάνει μια εξαιρετική δουλειά νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Απ' τη μία υπάρχουν τα αισθήματα, συναισθήματα και προσωπικές μνήμες. Πολύ σημαντικό, ανήκει στο πολιτιστικό κομμάτι, αλλά σε επίπεδο πολιτικό εμείς πρέπει να βασιστούμε στους επιστήμονες, οι οποίοι φεύγουν από το συναισθηματικό και μας επιτρέπουν να κάνουμε τις συζητήσεις αντικειμενικές. Αυτό που έχει σημασία στο δίκτυο κλειό Είχαμε τη δυνατότητα να τους συναντήσουμε στα πλαίσια της ευρωμεσογειακής διάσκεψης. Είναι τα λεγόμενα ε, διασταυρούμενα βλέμματα. Δηλαδή έχει σημασία να ξέρουμε όχι μόνο πώς βλέπουμε τους άλλους αλλά και πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Να ξέρουμε ακριβώς να δούμε το φασισμό με αυτόν τον τρόπο, να έχουμε και Ρώσους ιστορικούς, να έχουμε ε, Δυτικοευρωπαίους ιστορικούς, να συγκρίνουμε τις πηγές μας και τις αναλύσεις μας και να ξεφύγουμε από το συναισθηματικό. Φυσικά όμως και οι προσωπικές μνήμες και το συναισθηματικό είναι σημαντικές αλλά πρέπει να αποσυνδεθούν από την ιστορική μνήμη και δεν θα πρέπει να έχουν σχέση με την καθαρή επιστήμη. Λοιπόν κύριε Μιγκάλτσκι θέλετε να κλείσετε τη συζήτηση. Πέντε μαούνες. Ναι, θα ήθελα να λάβω το λόγο γιατί θα ήθελα να απαντήσω στις παρατηρήσεις. Καταρχάς, στον ε, κύριο Βάλε, Διβάλε. Πληθυντικό, είπατε. Ναι, βεβαίως. Ίσως δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για μία μόνο μνήμη, για δημιουργία μία μόνο μνημη Οι Πολωνοί, οι Γερμανοί, οι Βρετανοί μπορεί να έχουν διαφορετική μνήμη και ο στόχος ίσω αυτής της έκθεσης να είναι ακριβώς το να επισημάνει ότι υπάρχουν διαφορετικές ιστορικές μνήμε Και η δεύτερη παρατήρηση. Ολοκαύτωμα Γκούλαγκ. Ναι, δεν υπάρχουν θύματα πιο αξιοθρύνητα και λιγότερο αξιοθρύνητα, καλύτερα και χειρόμετρα, χιλιόχειρότερα. Δεν υπάρχει πιο αρεστός και λιγότερο αρεστός ολοκληρωτισμός, είτε πρόκειται για τους ναζί, είτε πρόκειται για τους κομμουνιστές. Εγκλήματα διέπραξαν, μπορούμε να κάνουμε διαφορετικές στατιστικές, αλλά όχι λογιστική στους, ε, στον των νεκρών. Τα θύματα των Γκούλακ ήταν θύματα όσο και αυτά του ολοκαυτώματο Και βεβαίως πάνω απ' όλα δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην αμνησία, στην λύθη να επικρατήσει. Γιατί έτσι ανοίγει και η πόρτα στον ε, εκδικητισμό, στην εκδικητικότητα. Για την κυρία Σάντσο Σμιτ ε, συμφωνώ με τη δική σας προσέγγιση ότι η Παιδαγωγική προσέγγιση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είμαστε ενήλικοι, έχουμε ιστορική γνώση και μνήμες. Η δουλειά μας όμως θα πρέπει να διαδοθεί, να εκλακιευθεί και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντική η παιδαγωγική προσέγγιση αυτής της διδασκαλίας. Επίσης δύο προσεγγίσεις σε σχέση με τον ναζισμό και τον κομμουνισμό, η διαδικότητα. Είναι απαράδεκτο αυτό που είπατε. Για τη διάσταση την οικονομική, τα οικονομικά. Ναι είναι χρήματα τα οποία επενδύονται τόσο καλά όσο και στο πρόγραμμα Έρασμους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει εδώ να επιδοθεί σε οικονομίες. Γιατί όποιο σπίτι χτίζεται πάνω σε σαθρά θεμέλια καταραίει. Αν λοιπόν πιστεύουμε ότι η μνήμη μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο του μέλλοντος, θα πρέπει σε αυτή να επενδύσουμε για την κυρία Τρίπελ που αναφέρθηκε σε διαφορετικούς ολοκληρωτισμούς. Ναι, ήταν διαφορετικοί οι αυτή αυτοί οι ολοκληρωτισμοί στην Ευρώπη, αλλά είχαν κοινά στοιχεία και πρέπει μέσα στην έκθεσή μας να τα επισημάνουμε. Συμφωνώ με την κυρία Τρίπελ. Είμαι πεπισμένος πως η Ευρώπη έχει προσφέρει το χειρότερο και το καλύτερο μαζί στον κόσμο. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση και χωρίς απαραίτητα να καταγράφεται στην έκθεση. Ξέρω ότι και πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει κάνει ό,τι καλύτερο και ό,τι χειρότερο στον κόσμο. Για την τελευταία συνάδελφο. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι απέχει τόσο πολύ δική σας εμπειρία από τη δική μου. Εγώ δεν είχα αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στην απεικιοκρατία γιατί δεν ανήκε ως εμπειρία στη δική μου γεωγραφική ζώνη. Θα το συζητήσω λοιπόν μαζί σας και διμερώς. Έχω κάθε διάθεση συνεργασίας μαζί σας. Η επικιοκρατία, χωρίς να είναι το ίδιο πράγμα με τον ναζισμό και τον ε, κομμουνισμό, που δολοφόνευσαν πολλούς ανθρώπους, οδήγησαν στο θάνατο πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι λοιπόν το ίδιο απαραίτητα με την απεικιοκρατία, αλλά θα ήθελα να μιλήσω με όλους εκείνους ε, οι οποίοι έχουν γνωρίσει από κοντά ίσως τα της απεικιοκρατίας. Θα προσπαθήσω λοιπόν να το συμπεριλάβω και όπως είπατε πρέπει να στηριχθούμε πάνω απ' όλα στη δουλειά των ιστορικών από την άλλη εμείς οι πολιτικοί είμαστε υποχρεωμένοι όπως λέμε να στηριχθούμε στη δουλειά των ιστορικών. Δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι ιστορικοί. Άρα ναι, πάνω σε κάτι θα πρέπει να στηριχθούμε, έστω και αν ξέρουμε ότι δεν συμφωνούν μεταξύ τους πάντα οι ιστορικοί. Ευχαριστώ πολύ. Από την Επιτροπή είναι ο κύριος Παύλ Τίχτελ εδώ. Είστε εδώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πήγες παρατηρήσεις για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες που αναφέρθηκε αρκετέ φορές και είναι ένα από τα κυριότερα, εάν όχι το κυριότερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να ενισχύσουμε την ιστορική μνήμη και στην Ευρώπη. Από το 2007 το 2013 έχει υποστηρίξει περίπου 300 προγράμματα και ήδη βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα, για προγράμματα ε, μνήμης. Θα ήθελα να σας δώσω μια εικόνα. Έχουμε λάβει περίπου 100 προγράμματα το 2007 και την τελευταία φορά που κάναμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος λάβαμε περίπου 400, βλέπετε την αύξηση. Ωστόσο ο προϋπολογισμός έχει παραμείνει περίπου ίδιος, θα έχουν αυξηθεί κατά λίγο τα κονδύλια, αλλά ε, αυτό οδηγεί ε, στο, στο να υπάρχουν προβλήματα με τον προϋπολογισμό. Από το 2014 έως 2020 η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο κανονισμό για το πρόγραμμα αυτό έχει προτείνει επίσης και την αύξηση του προϋπολογισμού ε, σε ποσοστία ε, κατά, ποσοστό για το πρόγραμμα από 4% σε 20%. Στόχος του προγράμματος θα είναι να εξετάσει ακριβώς την ευρωπαϊκή ιστορική μνήμη, αλλά επίσης και ε, δραστηριότητες μνήμης, για τα θύματα των ολοκληρωτικών καθεστώτων στην Ευρώπη. Η πρόταση του κανονισμού αναφέρεται στο ολοκαύτωμα, τον ναζισμό που οδήγησε στο ολοκαύτωμα, τον φασισμό, τον στο ελληνισμό και τον ολοκληρωτικό κομμουνισμό. Έχουμε όμως και μια διατύπωση η οποία αναφέρεται στα στιγμές εκείνες τις ιστορικές που διαμόρφωσαν την ευρωπαϊκή ιστορία και μέσω αυτής της διατύπωσης προσπαθούμε να καλύψουμε ιστορικά γεγονότα που διαμόρφωσαν ε, την ταυτότητα της Ευρώπης και την ιστορική της πορεία. Για παράδειγμα, εκεί θα μπορούσαμε να ε, συμπεριλάβουμε τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία ή επίσης τα... Ε, την πτώση του στίχου του 89 και τις επαναστάσεις στις διάφορες προενανατολικές χώρες και την επανένωση της Ευρώπης. Έτσι, θα μπορούσαμε να καλύψουμε και άλλες ιστορικές στιγμές της Ευρώπης που οδήγησαν στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Κάτι άλλο που επίσης συνδέεται με αυτά είναι η δυνατότητα να αναφερθούμε στις αξίες που μας συνδέουν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Το ζήτημα της απεικιοκρατίας, όπως είπα, δεν αναφέρεται στον κατάλογο των συγκεκριμένων ιστορικών γεγονότων όπως ο φασισμός, ο σταλινισμός, ε, ο κληρωτικό κομμουνισμός που αναφέρονται συγκεκριμένα στον κανονισμό, αλλά με την εναλλακτική αυτή διατύπωση ε, ζητημάτων ιστορικών γεγονότων που διαμόρφωσαν την Ευρώπη θα μπορούσαμε να καλύψουμε και την απεικιοκρατία. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε εδώ. Να συμμετάσχουν πολλοί φορείς γνώστες του ζητήματος. Χρειάζεται να υπάρξει ένας διάλογος με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών, των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα η Επιτροπή προσπαθεί να, να συνεργαστεί μάλλον με ιστορικούς, να εμπλακούν αυτοί στο διάλογο αλλά προσπαθούμε να αποφύγουμε να γίνει ένας απλός ακαδημαϊκός διάλογος μεταξύ ιστορικών. Θέλουμε αυτός ο διάλογος να ανοίξει στην ε, κοινωνία των πολιτών και στους Ευρωπαίους ε, πολίτες. Αυτό που προσπαθούμε να το επιτύχουμε μέσω του δικτύου ιστορικών κλειό. Τον Ιούνιο οργανώσαμε το ετήσιο συνέδριο του δικτύου κλειό που μας επέτρεψε να εξετάσουμε και τα προγράμματα που θα υποστηριχθούν από το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες τη συνέντευξη αυτή συμμετείχαν περίπου 200 εκπρόσωποι ε, ενώσεων καθηγητών. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαμε να απευθυνθούμε στους καθηγητές ιστορίας, όχι μόνο στις τοπικές αρχές. Γενικό, στόχος μας είναι να απευθυνθούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, σε όσο το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μπορούμε. Ωστόσο, οποιαδήποτε περικοπή υπάρξει στον προπολογισμό του προγράμματο. προφανώς θα επηρεάσει δυσμενώ τι πρωτοβουλίε και τα προγράμματα που θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μικάσκη. Δύσκολο το έργο σας. Ε, πολλές οι απαιτήσει που εκφράζονται από διάφορες πλευρές. Οπλιστείτε γερά. Το 2004 είχαμε μάλιστα μια ακρόαση εδώ με την οργάνωση Euroclio προσκεκλημένη. Μπορείτε να κοιτάξετε λοιπόν στα αρχεία μας. Και εκεί θα βρείτε υλικό. Βεβαίω το ε, προσωπικό της γραμματείας να σας βοηθήσει. Δεν είναι και τόσο παλιά το 2004. Θα βρείτε ίσως υλικό εκεί που μπορεί να σας χρησιμεύσει σαν βάση. Και για να ανατέκρουστε αυτά σε αυτά που είπατε και εσείς και η Επιτροπή, πρέπει να πω ότι αισθάνομαι μια θλίψη, διότι όταν λέτε να γίνουν αυξήσεις, πού θα γίνουν αυξήσεις, κατά 23% περικόπτεται το πρόγραμμα. Ε, δεν βελτιώνεται σε τίποτα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε λοιπόν να επικροτήσουμε την Επιτροπή σε αυτή την περικοπή της. Και περικόπτεται το μεγαλύτερο, κατά το μεγαλύτερο τμήμα στον τομέα αυτόν. που όσο και αν μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτό ο τομέα, κάποιοι άλλοι θα πρέπει να περικοπούν. Η αδελφοποίησης ε, πόλεων, παραδείγματι, που έχουν πολύ, καλό, πολύ καλές επιδόσεις στο learning by doing. Όλα αυτά ξέρουμε ότι θα δουν περικοπές. Δεν βοηθάει σε τίποτα αυτό που κάνετε να περικόπτετε τον προϋπολογισμό. Ξέρω ότι θα... Ε, κάνετε ό,τι μπορείτε. Βλέπω από το πρόσωπό σας ότι κάνετε φιλότιμες προσπάθειες, αλλά δεν μπορεί να δουλεύει έτσι η Επιτροπή. Ήδη υπάρχει μια αυτοπερικοπή, ένας αυτοπεριορισμός κατά 5%. Και τώρα προσθέτει άλλο ένα 19%. Είναι όνειδος, όνειδος και για το κοινό μας εγχείρημα. Και ε, εάν μπορέσει αυτή η έκθεση του κυρίου Μιγκάλσκι να αναδέψει λίγο τα νερά στην Επιτροπή και να κάνει κάποιους να ξανασκεφτούν αυτές τις περικοπές, τότε ίσως να κερδίσουμε κάτι και ίσως και οι συνάδελφοι που διαπραγματεύονται το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο να κάνουν μια προσπάθεια παραπάνω. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία, καλό καλοκαίρι. Μέχρι το φθινόπωρο έχετε χρόνο για να καταθέσετε την έκθεση σας κύριε Μιγάλσκι. Θα είναι δύσκολο να εξισορροπήσετε όλες τις απόψεις. Ε, είσαστε πάνω σε ένα πολύ λεπτό στρώμα πάγου Πολλοί είναι οι υποτιθέμενοι ιστορικοί εδώ στην αίθουσα και γύρω από την αίθουσα που θα έχουν τις επόψεις τους να εκφράσουν. Και εγώ που έχω την οπτική της δύση στην υπόθεση αυτή, πρέπει να πω ότι το 2004 όταν ενταχθήκατε όλοι εσείς, όλες εσείς στα κράτη, δυσκολευτήκαμε με, τις, ε, με τους εορτασμούς του 2005 να καταγράψουμε τοποθετήσεις που να εκφράζουν σωστά τις θέσεις της δικές σας αυτών των κρατών που από το 1945 και μέχρι εκείνη την ώρα, μέχρι το 2004, βρίσκονταν από την άλλη πλευρά και που δεν είχαμε λάβει υπόψη ποτέ και που δεν γνωρίζαμε τι σημαίνει για αυτούς ο εορτασμός των ε, 60 χρόνων από το τέλος του πολέμου το 2005. Γι' αυτό λοιπόν χρειάστηκε να κοιτάξουμε με διαφορετική ματιά να δούμε τα δικά σας, τα δικά σας επιχειρήματα. Πολλά είχαμε λοιπόν να μάθουμε, τα μάθαμε πιστεύω. Και είμαι βέβαιο ότι και η δική σα έκθεση θα είναι μια πολύ καλή έκθεση. Σα εύχομαι κάθε επιτυχία. Στι 17 Σεπτεμβρίου θα έχουμε πιστεύω την χαρά να απολαύσουμε την πρώτη σας έκθεση. Ε, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ ενδιαφέρον βρήκα το ότι αυτό που είπατε ότι κάποιοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχουν ενστερνιστεί πολύ σοβαρά αυτή την υπόθεση. Και αν σκεφτούμε ότι και στη Γερμανία καλά καλά δεν ξέρουν πλέον ε, οι νέοι τι συνέβαινε πριν από 20 χρόνια. Υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν ε, τι συνέβαινε στην Ανατολική Γερμανία, πρώην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και τι συνέβαινε στη Δυτική. Έχουμε πολλή δουλειά λοιπόν να κάνουμε στην ιστορία, πολλή πράγματα να εξηγήσουμε στα παιδιά. Ιδάλλως, εάν δεν έχει πια αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ιστορία, δεν θα έχει και μέλλον. Και χαίρομαι που έχετε αναλάβει την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ και τώρα πάω στο σημείο 4, όχι στο 5 της ημερησίας εντάξεως. Έχουμε προσκαλέσει. Έχω αναθέσει μάλλον στην ομάδα μελέτης το καθήκον να κάνει μια παρουσίαση. Ουνιβερσιτά Πολυτέχνικα de Madrid, τον κύριο Κλάουδιο Φέιο συγκεκριμένα και την κυρία Ελίσσα Τελανούε Σάντσες Κασκάδο. Τους καλώ να έρθουν εδώ να μας κάνουν την παρουσίασή τους για το δημόσια και εμπορικά μοντέλα στην ψηφιακή εποχή. Α Ας μην συνεχίσω εγώ με τη διάλεξή μου. Ας παρακαλέσω τους ε, ερευνητέ μας να έρθουν να μας κάνουν την παρουσίαση. So, Who is beginning? Mr. Claudio Okay. ξεκινάει ο κύριος Φέιο Παρακαλώ τώρα να μας ακούσει λίγο το προσωπικό εδώ. Okay, you have the floor. Έχετε το λόγο. Τι θα μιλήσετε. Α, η Αγγλικούλια, ωραία. Okay. Um, first of all, good afternoon everybody. It is uh, truly a pleasure to be here. Με χαρά είμαι ανάμεσά σας. Πιστεύω πραγματικά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, Πρόεδρε. Είμαι ο συντονιστής της συγκεκριμένης μελέτης, αλλά έχω μαζί μου εδώ έναν συνάδελφο που έχει εργαστεί και πιο πίσω. Έχουμε και την κυρία Ντελανουέζ που είναι διευθύντρια, αν θέλετε, της εταιρεία η οποία ασχολήθηκε με την διαμόρφωση αυτής της πρότασης. Ε, παρουσιάζουμε ένα πραγματικά απλό storyline, δηλαδή μια επισκόπηση των στόχων της εμβέλειας, και θα εξηγήσουμε επίσης ε, και ό,τι έχει σχέση με το περιεχόμενο των βιομηχανιών των μέσων και επίσης θα σταθώ στο λεγόμενο δημόσιο περιεχόμενο έτσι ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε ακριβώς ποια είναι, το ποιο είναι τα, τα σημαντικά σημεία. Cultural creative content is digitally delivered to and accessed by the wider public in Europe, so the essence of the report is in the digitally delivered. Η ουσία είναι ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται οι πληροφορίες μέσω ακριβώς των συγκεκριμένων τρόπων και μέσων. αν μπορεί κανείς να βγάλει κάποια συμπεράσματα από τη χρήση του δημοσίου περιεχομένου σε σχέση με το επιχειρηματικό εμπορικό περιεχόμενο, βλέπει ακριβώς τι γίνεται σε διάφορους τομείς όπως σε εφημερίδες, αν και υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι δεν είναι πολύ πιο προχωρημένοι στη μετάδοσή τους και στα μέσα μετάδοσης όπως η μουσική.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 η δομή αυτή διαιρείται σε τρεις φάσεις. Από τη μία έχουμε την παραγωγή, την διανομή και την κατανάλωση. Και έχουμε και αποφάσεις οι οποίες αφορούν και τα τρία αυτά στάδια. Το κόστος της διανομής με το διαδίκτυο προφανώς έχει μειωθεί πάρα πολύ Έχει αυξηθεί βέβαια το κόστος της παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανείς με τις ίδιες επενδύσεις να επιδιώξει υψηλότερη ποιότητα ή και να μεταβεί εκτός της παραδοσιακής σφαίρας παραγωγής. Και τελικά έχει αλλάξει και η χρήση του τρόπου κατανάλωσης και πώς συνδέεται ο τρόπος της χρήσης με το περιεχόμενο του μέσου. Έχουν υπάρξει λοιπόν οικονομικές αλλαγές, έχουν υπάρξει αλλαγές κοινωνικο-οικονομικές και αυτά επηρεάζουν τον τρόπο της παραγωγής. Υπάρχει το θέμα της παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και η παραδοσιακή βιομηχανία των μέσων άργησε λίγο να αντιδράσει, αντέδρασε μειοπικά θα έλεγα σχετικά με τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν. Μπράβο. Μπράβο. So in fact the decision is not completed, no? There's still some problems as as obvious. Okay. So so I was I was saying um let's say that this behavior this approach of the traditional industry Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε όπως είπα η βιομηχανία δεν ήταν ο καλύτερος και προκάλεσε καθυστερήσεις στο πώς μπόρεσαν και νέοι πρωταγωνιστές να ενταχθούν στον συγκεκριμένο χώρο. Για να τελειώσω λοιπόν την περιγραφή της κατάστασης όπως έχει σήμερα, έχουμε και κάποιους νέους παίκτες αν θέλετε, υπήρξε μια άμεση σχέση ανάμεσα στους παραγωγούς από τη μία και τους καταναλωτές από την άλλη. Σιγά σιγά βέβαια η έννοια της διαμεσολάβησης άρχισε να παίρνει μεγαλύτερο βάρος, η έννοια των νέων ενδιαμέσων θα τους ονομάσω. Και πέραν αυτού θα πω ότι οι παραδοσιακές ε, δραστηριότητες που υπήρχαν στο παρελθόν εξακολουθούν να επηρεάζουν τα πράγματα τα λεγόμενα legacy features. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουν ακόμα και αυτοί οι παραδοσιακοί διανομής μέσων να μπορέσουν να βρουν θετικούς τρόπους έτσι ώστε να δημιουργηθεί προστιθέμενη οικονομική και κοινωνική αξία μέσα από τα προϊόντα τα οποία μεταδίδουν. Τώρα, πώς έχει διαμορφωθεί το τοπίο μετά από τις τελευταίες βίαιες αλλαγές. Τώρα έχουμε αρχίσει να έχουμε μία πρώτη εικόνα του πώς θα πάνε τα πράγματα στο μέλλον. Γνωρίζουμε ότι οι παραδοσιακές βιομηχανίες θα σμικρίνουν ακόμα περισσότερο ιδιαίτερα στον τομέα της μουσικής. Φαίνεται βέβαια ότι στον τομέα της μουσικής οι παραδοσιακές δραστηριότητες έπεσαν αρκετά και τώρα από εδώ και πέρα έχουν αρχίσει και προσαρμόζονται. Έχουμε νέους παίκτες, έχουμε νέες μορφές κυριαρχίας της αγοράς με διαφορετικές αξίες, όχι πολιτιστικές αλλά διαφορετικές αξίες. Άλλες καλές, άλλες κακές. Το παραδοσιακό μοντέλο σαν παράδειγμα μπορεί να απολύει στη συγκεκριμένη φάση προϊόντα ηλεκτρονικά ή ηλεκτρολογικά αλλά αυτό έχει αρχίσει ε, να είναι στο ίδιο επίπεδο σημασίας με το περιεχόμενο των μέσων τα οποία οι μηχανισμοί αυτοί καλούνται να μεταδώσουν. Και τίθεται και στην περίπτωση του περιεχομένου το πρόβλημα που ίσχυε και στις περιπτώσεις ε, ε, των παραδοσιακών ηλεκτρονικών βιομηχανιών, δηλαδή συνεργασίες, δημιουργία οικοσυστημάτων, προσπάθειες επικυριαρχίας των προϊόντων αυτών, της αγοράς των προϊόντων αυτών, κοινέ πλατφόρμες, προστασία από hacking. Όλα αυτά είναι τμήμα θα έλεγα των δομών αυτής της νέας ε, πλευράς της βιομηχανίας των μέσων. Έχουμε επίσης διαφορές και στην παραγωγή και στην διανομή και στην ε, κατανάλωση. Έχουμε στο επίπεδο της παραγωγής ε, αυτό που ονομάζουμε διασταυρούμενη εμπειρία μέσων. Έχουμε τη συνεργασία πολλών μέσων που καταλήγουν σε ένα προϊόν. Έχουμε επίσης χαμηλότερα εμπόδια για να μπουν στην αγορά κάποιοι φορείς από ό,τι στο παρελθόν. Έχουμε την δυνατότητα ακόμα και για διανομή και παραγωγή μη επαγγελματιών στον συγκεκριμένο χώρο που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Στον τομέα της διανομής αναφέρθηκα στα λεγόμενά μου, αναφέρθηκα μάλλον ε, και στα θέματα των ενδιαμέσων οι καταναλωτές λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, έχουμε πάρα πολλά είδη μέσων, προσωπικά, συλλογικά, κοινωνικά, ιδιωτικά, επιχειρηματικά Έχει πάρει λοιπόν μια νέα μορφή η συγκεκριμένη αυτή βιομηχανική οικονομική δραστηριότητα. Έχουμε και τα λεγόμενα business models. Έχουμε σαν βασικό χαρακτηριστικό εδώ την έλλειψη σημασίας της έννοιας των συνόρων, του εδάφους της παραγωγής. και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα σε επίπεδο ρυθμίσεων και διακανονισμού γιατί προηγουμένως η παραγωγή και η διανομή και η κατανάλωση ήταν κάτι το οποίο ρυθμίζεται μέσω των εθνικών ε, ρυθμίσεων και αρχών. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Υπάρχουν τρία επιχειρηματικά μοντέλα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε τις διαφημίσεις οι οποίες περνούν και στα λεγόμενα κοινωνικά μέσα ε, ε, δικτύωσης, στη συλλογή πληροφοριών για τους καταναλωτές ήταν κάτι το οποίο δεν έκαναν στο παρελθόν τα παραδοσιακά μέσα, τα οποία στόχευαν γενικά μεγάλο κοινό. Έχουμε επίσης τα νέα αυτά πρότυπα το πέρασμα από ένα συγκεκριμένο προϊόν σε μια υπηρεσία περισσότερο. Και τέλος, σε ορισμένους τομείς βλέπουμε και κάποια επιμέρους νέα πρότυπα παραγωγής που ισχύουν για τον συγκεκριμένο τομέα. Τα clouds και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτές είναι οι ιδέες γενικά ε, σχετικά με την κατάσταση που βρίσκεται ο συγκεκριμένος τομέας. Μιλάμε για ένα ετερογενές περιβάλλον, υπάρχουν όπως είπαμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ανατομέα. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αγορά κυριαρχείται από τις Ηνωμένε Πολιτείες, αν και υπάρχουν σε εθνικά επίπεδα και κάποια εθνικά χαρακτηριστικά πολύ σοβαρά. Οι βασικές προκλήσεις είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και σε επίπεδο κινηματογραφικό και σε επίπεδο προβολή σε αίθουσες δηλαδή των κινηματογραφικών έργων και σε επίπεδο διανομής με DVD και σε επίπεδο πληρωμής ένα έργο μέσω τηλεόρασης. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές αλλαγές εδώ που έχουν συμβεί και δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι τα πρότυπα που θα επιβιώσουν μελλοντικά. Υπάρχει μια κάποια σύγχυση. Υπάρχει επίσης ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με το πώς μπορούν να προβάλλονται κάποιες ταινίες σε διαφορετικές περιοχές λόγω των περιορισμών ε, για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Έχουμε επίσης και την διανομή και κατανάλωση ψηφιακή κινηματογραφικών έργων που είναι ιδιαίτερα περιορισμένη ακόμα βέβαια. Έχουμε κάποια στοιχεία σχετικά όχι πρόσφατα. Οι στατιστικές ε, καθυστερούν <clears throat> αλλά εν πάση περιπτώσει τα ποσοστά κάποτε γύρω από, το online, από την online διανομή ήταν χαμηλά. Τώρα για την ψηφιοποίηση του κινηματογραφικού προϊόντος. Αυτό μειώνει κόστος, απλοποιεί την επεξεργασία της παραγωγής και επιτρέπει την εφαρμογή καινοτόμων, επιχειρηματικών επιχειρηματικών προτύπων. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ενδιαφέροντα, πολλές ενδιαφέρουσες εμπειρίες οι οποίες καλύπτουν κάποιους από τους τομείς που προανέφερα. Αυτό φαίνεται γιατί έχουμε εδώ έναν τομέα σαν παράδειγμα που είναι πολύ σημαντικός για την ψηφιακή διανομή των προϊόντων. Έχουν επίσης στο επίπεδο ελέγχου των πνευματικών δικαιωμάτων αρκετά ισχυρή θέση οι παραγωγοί οι Ευρωπαίοι. Έχουν πολλές επίσης ευρωπαϊκές καινοτομίες σε παιχνίδια ε, μέσω διαδικτύου. Έχουμε λοιπόν διάφορα επιχειρηματικά πρότυπα νέου τύπου και εδώ. Έχουμε επίσης μοντέλα που καθορίζονται από τη δυνατότητα πρόσβασης είτε μέσω του browser είτε μέσω ε, μια συγκεκριμένης εφαρμογής που έχει προαγοράσει ο πελάτης είτε μέσω του κινητού μέσου αναπαραγωγής. Έχουμε διαφορετικά πρότυπα για την πληρωμή πληρωμή αναφόρτωση, έχουμε την επαναλαμβανόμενη σύνδρομη, έχουμε την πληρωμή για τις προεκτάσεις, τα προεκτάματα των παιχνιδιών, ε, έχουμε επίσης ε, και τις λεγόμενες κονσόλες, ε, τα τηλέφωνα, τους υπολογιστές, τα tablets κτλ. Και έχουμε επίσης και το λεγόμενο μοντέλο freemium που είναι κάποια βασικά χαρακτηριστικά δωρεάν. Τώρα, τα βιβλία. Στα πλαίσια αυτών των αγορών που μας ενδιαφέρουν τα βιβλία στην διαδικασία της ψηφιοποιημένης αγοράς ήρθανε με μεγάλη καθυστέρηση. Το 2012 τα ηλεκτρονικά βιβλία ήταν μόνο το 4,5% των συνολικών πωλήσεων στις, αναπτυσσόμενες, ή στις αναπτυγμένες χώρες. Ήταν χαμηλό ποσοστό εν πάση περιπτώσει. Είναι η μόνη αγορά όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι κυρίαρχες αλλά δυστυχώς οι αμερικανικές επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες ελέγχουν τη μετάβαση στην ψηφιοποίηση, στην ψηφιακή ε, βιομηχανία. Τώρα υπάρχουν νέα επιχειρηματικά πρότυπα στα οποία έχουμε καθυστερήσει. Εμείς ε, ε, στην ουσία την αγορά του χαρτιού την μεταφέρουμε στον ψηφιακό κόσμο. Έχουμε όμως πολύ περισσότερες δυνατότητες τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Υπάρχουν τα κλειστά πρότυπα που συνδέονται με συγκεκριμένους αναπαραγωγείς που δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς τη χρήση τους κάνουν μία συγκεκριμένη δουλειά και συνδέονται με μία συγκεκριμένη πλατφόρμα ανάγνωσης βιβλίων στη συγκεκριμένη περίπτωση και έχουμε επίσης και τα ανοιχτά πρότυπα που βασίζονται σε πλατφόρμες online όπως περιοδικά, εφημερίδες και εκεί έχουμε αύξηση των συνδρομών, έχουμε αύξηση των εσόδων των εφημερίδων και των περιοδικών. Βλέπουμε να υπάρχει μια έκρηξη επίσης των online ειδήσεων Φαίνεται ότι υπάρχει ζήτηση αλλά η βιομηχανία δεν είναι σε θέση να καλύψει τη ζήτηση αυτή γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με το ίδιο είδος της δημοσιογραφίας που απαιτείται στο γραπτό κομμάτι με το ψηφιακό κομμάτι. Υπάρχει επίσης και ένα ποσοστό δοκιμαστικών ρυθμίσεων, ε, ε, κάποιες ε, δυνατότητες που υπήρχαν και δοκιμάστηκαν απέτυχαν και ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει τα πράγματα και δεν έχουν επιλεγεί τα μοντέλα σύμφωνα με τα οποία κάποιος προσθέτει στο βασικό χαρακτηριστικό το, μεταφερόμενο στοιχείο κάποια επιπλέον στοιχεία τα οποία κοστίζουν επιπλέον επίσης. Παρουσίασα πολύ συνοπτικά λοιπόν τον τρόπο λειτουργίας του εμπορικού τομέα και τώρα να μιλήσω για το δημόσιο περιεχόμενο ε, και τους δημόσιους ιστοτόπους. Η βασική ιδέα είναι ότι υπάρχουν διαφορετικοί, ε, διαφορετικά έργα τα οποία μεταφέρονται σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε έργα τα οποία είναι ήδη ελεύθερης χρήσης, έχουμε έργα τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και έχουμε και μια τρίτη κατηγορία όπου τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε ένα ιδιωτικό τομέα αλλά κατέχονται από το δημόσιο. Τα λεγόμενα ορφανά έργα και τα έργα τα οποία δεν είναι πλέον σε επίπεδο εμπορίας στη συγκεκριμένη φάση. Αυτός είναι ένας τομέας ο οποίος ακόμα είναι αρκετά πίσω σε επίπεδο ψηφιοποίησης. Μόνο το 6% του ευρωπαϊκού πολιτιστικού περιεχομένου είναι προσβάσιμο σε ψηφιακό τρόπο, online. και αν θέλουμε να μιλήσουμε και για διαδραστικές δυνατότητες επικοινωνίας online, τότε το ποσοστό είναι ακόμα πιο χαμηλό. Λοιπόν, η διαδικασία της δημιουργίας λοιπόν ψηφιακού περιεχομένου σε δημόσιο επίπεδο ε, μέχρι τώρα έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά. Καταρχάς έχει υπάρξει προσοχή στην ίδια τη διαδικασία της ψηφιοποίησης και αυτό είναι πρόβλημα γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι μόνο της προσπάθειας που πρέπει να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό το να γίνει αυτό βέβαια, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και το καθεστώς σε επίπεδο πνευματικών δικαιωμάτων, είναι προφανές, και θα πρέπει επίσης και η διάθεση online των προϊόντων αυτών να είναι δεδομένη και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα. Είναι μια πολυδιάσπαση, διαπιστώνουμε μια πολυδιάσπαση της ψηφιακής αγοράς δημοσίου περιεχομένου αποτελείται από ορισμένα προγράμματα βραχυπρόθεσμα κυρίως και επίσης οι βασικές μορφές χρηματοδότησης είναι το δημόσιο με πολύ μικρή συμμετοχή σταθερής ιδιωτικής χρηματοδότησης. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά εμπόδια στον τομέα του δημοσίου περιεχομένου Έχουμε έλλειψη χρηματοδότησης, έχουμε ξεκάθαρες αποδόσεις, έχουμε υψηλό κόστος ψηφιοποίησης, έχουμε ανώριμα επιχειρηματικά πρότυπα, δεν υπάρχουν οδικοί χάρτες, υπάρχει έλλειψη συντονισμού, υπάρχει έλλειψη οικονομιών κλίμακας, υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων στο εσωτερικό των δημοσίων υπηρεσιών, και υπάρχει επίσης και έλλειψη διαπραγματευτικής δυνότητας όπως και έλλειψη συνειδητοποίησης <coughs> του προϊόντος από τους χρήστες. Από την άλλη υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες, υπάρχει ένα συγκεκριμένο δυναμικό, υπάρχει υψηλή ζήτηση η οποία πρέπει να ικανοποιηθεί ανάλογα. Υπάρχουν πολλά που μένει να γίνουν λοιπόν. Τελειώνοντας λοιπόν Φτάνω στο τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης και έχουμε διορθώσει τις ιδέες που είχαμε. Έχουμε συλλέξει μάλλον πέντε βασικές ομάδες συστάσεων. Βασικά. Και θα σας το παρουσιάσω με τον πιο απλό δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να κατανοήσετε το μήνυμα αυτής της προσπάθειας. υπάρχει ανάγκη για περισσότερη χρηματοδότηση. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η καιρή, αλλά αυτό εξηγείται ε, από τις εξωτερικές αποδόσεις που είναι πάρα πολύ θετικές. Πρόκειται για μία δηλαδή οικονομική προσπάθεια που βελτιώνει πολλές άλλες δυνατότητες οικονομικές για την κοινωνία. Θα απαιτηθούν λοιπόν ε, ε, μορφές χρηματοδότησης, τις διασταυρούμενες μορφές παραγωγής, σε προγράμματα και σε μέσα για καινοτόμους επιχειρηματίες, θα πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι για τη χρήση του περιεχομένου, θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες νέες πλατφόρμες ευρωπαϊκού επίπεδου και ευρωπαϊκών οικοσύστημάτων, το μίσο όπου έτσι και αλλιώς είμαστε μπροστά, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα διαμεθοριακής διανομής, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και για το δημόσιο περιεχόμενο και θα πρέπει να υπάρξει προσπάθεια αποφυγής των αποκτών επικαλύψεων. Ε, αυτός είναι ο πρώτος τομέας των συστάσεων. Ο δεύτερος τομέας είναι η καλύτερη μορφή συντονισμού και να μειωθεί το κόστος των συναλλαγών το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό σήμερα έτσι ώστε να επιτρέψει να αναπτυχθεί κάτι από ένα κράτος μέλος και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη και να διευρυνθεί η χρήση των επιχειρηματικών προτύπων σε όλες τις χώρες. Πρέπει να υπάρξει συντονισμός των δράσεων, πρέπει να υπάρξει περιεχόμενο επιπλέον στις υπάρχουστες πλατφόρμες και πρέπει να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών απέναντι στους παροχείς. Δηλαδή να αποφύγουμε παραβιάσεις και προβλήματα απάτες κτλ τρίτος ε, θα έλεγα, τρίτος, τρίτο σύνολο των συστάσεων είναι ότι απαιτείται φυσικά μια βελτίωση της έκδοσης αδειών, της αδειοδότησης ε, σε διεθνές επίπεδο ε, του καθεστώτος πνευματικής προστασίας, πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός των μορφών των ισχυουσών αδειών θα πρέπει επίσης να υπάρξει ίσως κάτι που να ονομάζεται Ευρωπαϊκή Άδεια Κυκλοφορίας έργου. Θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και εφόσον ισχύει σε μια χώρα να μπορεί να ισχύσει και σε άλλες χώρες κάτι το οποίο θα αυξήσει την δυνατότητα διανομής περαιτέρω του προϊόντος. Θα πρέπει επίσης να ανοιχνεύσουμε την έρευνα και να προωθήσουμε και νέους τρόπους παροχής δημοσίου περιεχομένου. Υπάρχουν δυνατότητες καινοτομίας, μπορώ να σας δώσω και άλλα παραδείγματα. Υπάρχει τρόπος δηλαδή. Δεν είναι όλα ολοκληρωμένα τώρα. Ε, τέταρτο θα έλεγα σύνολο συστάσεων είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο δημόσιο περιεχόμενο, η αξιολόγηση της άμεσης παροχής του περιεχομένου, η κοινωνική καινοτομία στην διανομή του, του περιεχομένου, η δημιουργία ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων σχετικά με το δημόσιο περιεχόμενο, νέα πρότυπα, τα λεγόμενα freemium, και επίσης καινοτόμες εμπειρίες των χρηστών, ε, ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα και φτάνω στο τελευταίο κομμάτι των συστάσεων, υψηλού επίπεδου ικανότητες των επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διανομή του δημοσίου, ε, των δημοσίων μέσων. Σας ευχαριστώ πολύ. το βαρύ το πιάτο που μας σερβίρατε. Με ακούτε. Στην αρχή μπορώ να πω ότι δεν μπορούσα να παρακολουθήσω ακριβώς. Στο τέλος κάπου ξαναβρήκα τα νερά μου. Το τέταρτο σημείο είναι αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η εκπαίδευση και βέβαια με το αναλυτικό πρόγραμμα αναφέρεστε σε κάτι στο οποίο ίσως δεν είναι τόσο εύκολο να υλοποιηθεί. Άλλα χρόνια τώρα προσπαθούμε να εξηγήσουμε στα κράτη ότι χωρίς ε, γνώσεις και δεξιότητες χρήσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Μας ε, περιγράψατε λοιπόν μια εικόνα με όλες αυτές τις νέες δυνατότητες που προσφέρετε. Οφείλω να πω όταν βαρύ το πιάτο και έτσι θα πρέπει να πάρω κάποιο χρόνο για να το χωνέψω. Αλλά ίσως κάποιοι συνάδελφοι είναι έτοιμοι να τυπώσουν τις ερωτήσεις τους χωρίς απαραίτητα να εμβαθύνουμε. Κυρία Μπένερα Καταρχάς θα ήθελα να έξω τις ευχαριστίες μου, ήταν πολύ σαφής η σύνθεση, παραμένει όμως σύνθεση. Δύο σημεία. Στις συστάσεις σας μιλάτε για τη σημασία της χρηματοδότησης, την ανάγκη εξεύρωσης χρηματοδότησης. Στα κοινωνικά δίκτυα τη χρηματοδότηση την εξασφαλίζει η διαφήμιση. Άρα πρόκειται για μια παράλληλη χρηματοδότηση, γιατί μπορεί να είναι επισήμω ε, δωρεάν η χρήση των μέσων, αλλά ακολουθείται από ε, διαφημίσεις. Θεωρείτε λοιπόν ότι η διαφήμιση ως μέσο χρηματοδότησης περιεχομένου και ψηφιακού υλικού ε, είναι κάτι το σκόπιμο. Εγώ ανησυχώ λίγο γι' αυτό. Αλλά δεν θέλω να δω τις απαντήσεις σας. Και εάν υπάρξει αυτή η παράλληλη χρηματοδότηση, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει πρόσφατα σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις Google κτλ. Αυτό της φορολογίας που επίσης αποτελεί μέσον χρηματοδότησης. Έχετε σε αυτό συστάσεις και με τι μέσα μόχλεψης μπορείτε να εξασφαλίσετε αυτή τη χρηματοδότηση. Σε ένα κόσμο τόσο περίπλοκο, σε ένα κόσμο που δεν γνωρίζει ε, εθνικά σύνορα, η υλικά όρια και που σχετίζεται τόσο πολύ με τις υπηρεσίες. Άιρο κόσμο. Πώς μπορεί δηλαδή να εξασφαλιστεί η φορολόγηση εφόσον είναι σκόπιμο αυτών των, ε, αυτών των υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Για απάντηση. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω με την πρώτη, με τη δεύτερη, για τη φορολογία. Θα θυμίσω λοιπόν μια ταινία όπου ο πρωταγωνιστής κάποια στιγμή έχει, την ατάκα μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Ε, θα μιλήσω λοιπόν και εγώ ελεύθερα. Υπάρχει λοιπόν η έννοια αυτή του ανταγωνισμού του φορολογικού μεταξύ κρατών μελών που είναι μια πολύ λάθος ιδέα. Και έχοντας ε, σπουδές ε, οικονομολόγου μπορώ να σας πω με αυτή την ιδιότητα ότι εάν προσφέρεται μια υπηρεσία για την κοινωνία, μπορούν ωραιότατα να ε, ζητηθούν και οι σχετικοί φόροι. Αυτό έχω να πω για τη φορολογία. Για την πρώτη ερώτηση και τη σημασία της χρηματοδότησης. Πρέπει καταρχάς να γίνει μια διάκριση μεταξύ εμπορικού και δημοσίου περιεχομένου. Όταν μιλούμε για δημόσιο περιεχόμενο, σε μια τέτοια εποχή όπως αυτή της οικονομικής κρίσης που διαβιώνουμε, σημαίνει ουσιαστικά ε, τη δυνατότητα για εισαγωγή μιας εταιρική σχέσης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μιας ΣΔΙΤ. Αυτή θα ήταν η μόνη λύση που θα έβρισκα. Θα έπρεπε δηλαδή ο δημόσιος ε, χώρος να αφήσει περιθώριο για την δραστηριοποίηση του ιδιωτικού, ώστε να λειτουργήσει μια τέτοια σχέση. Είναι το μόνο που θα βλέπω αυτή τη στιγμή. Για το εμπορικό περιεχόμενο, ίσως υπάρχει μια υπερβολική αντίδραση ως προς την ε, διαφήμιση, μια υπερβολική, ένας υπερβολικός ενθουσιασμός για την ε, διαφήμιση. Όλοι θεωρούν ότι τα πάντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τη διαφήμιση, αλλά δεν μπορεί να τα λύσει όλα τα προβλήματα η διαφήμιση, καθώς ε, μάλιστα απαιτεί και χρήση προσωπικών δεδομένων μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται κάτι το οποίο να μας εξασφαλίζει πλήρη κατανόηση αυτής της κατάστασης. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με διαφήμιση κάθε τύπου περιεχόμενος εκ τούτου. Ένας τρόπος θα μπορούσε να είναι και πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα προκειμένου είναι η ε, μουσική. Ε, θα μπορούσε να είναι λοιπόν η ε, συνδρομή, ψηφιακή συνδρομή που θα μπορούσε να πάρει διάφορου τύπου. είτε ψηφιακή συνδρομή μόνο για μία μέρα, είτε ψηφιακή συνδρομή μόνο για συγκεκριμένο είδο μουσικής, διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, που θα ήταν κάτι διαφορετικό από την διαφήμιση. Και αυτή είναι η δική μου άποψη στην έκθεση αυτή. Η Πρόεδρος. Βλέπω ότι είστε λίγο πολύ ικανοποιημένοι με την απάντηση. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν. Ε? Μάλικα. Ναι, σχετικά με τη χρηματοδότηση του πνευματικού, της πνευματικής παραγωγής, πρόκειται εδώ για ένα μεγάλο ε, ζήτημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα ως Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτούμε την πνευματική παραγωγή των, των καλλιτεχνών μας. Μια επιχειρηματολογία που προχωρεί και δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι ε, ποια είναι η ορολογία που χρησιμοποιείται. Ε, θα ήταν όμως ε, αυτή της σε μικρή έκταση, με μικρά ποσά χρηματοδότησης από πολλούς χρήστες αυτής της παραγωγής. Δηλαδή μικρά ποσά τα οποία χρησιμοποιούνται τελικά για να χρηματοδοτηθεί, για να συντηρηθεί αυτή η πνευματική παραγωγή. Ναι, στην έκθεση αναφερόμαστε στην κοινωνική καινοτομία σε αυτό θα θέλαμε να αναφερθούμε για τα αισθήματα της χρηματοδότησης. Προσωπική μου έποψη είναι ότι και είναι ενδιαφέρον, ενδιαφέρουσα λύση, αλλά και ε, υπερθυμημένη σε έναν βαθμό. γιατί όλοι στρέφονται μαζικά προς την ίδια κατεύθυνση. Αλλά όπως είπα, καλό θα είναι να ευαισθητοποιηθεί ο καταναλωτής ως προς τη σημασία του δημόσιου αγαθού για να εμπλακεί. Τώρα θέλουμε την κοινωνική κοινοτομία να την βάλουμε μέσα στην ε, κοινωνική χρηματοδότηση. Είναι ευρύτερο βέβαια το θέμα της κοινωνικής ε, καινοτομίας από αυτό της της κοινωνικής χρηματοδότησης, αλλά πάντως υπάρχει μια σχέση. Και πάλι επαναλαμβάνω, είναι ίσως υπερβολικός ο ενθουσιασμός που εκφράζεται. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Δεν βλέπω να στείλει κανείς άλλος το λόγο για να διατυπώσει ερωτήσει προς τον ομιλητή. Θα τα λάβουμε όλα αυτά που είπατε υπόψη. Το έγγραφό σας μας ε, δίνει υλικό και νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον και για άλλες επιτροπές, ε, όσες είναι αρμόδιες για το περιεχόμενο περισσότερο. Και καλό θα ήταν να διαβιβάσουμε. Να μπορέσουν και οι να να λάβουν γνώση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φεϊού και η κυρία Ελίζα έστησε Σιάντσες Κασκάδο, η οποία καθόταν εδώ πίσω και όχι μπροστά. Δεν ε, ξέρω ότι ήσασταν εδώ, δεν σας γνώρισα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κατόπιν τούτου ολοκληρώσαμε την δημόσια συνεδρίασή μας. Τώρα θα συνεχίσουμε με τους συντονιστές, αλλά περιμένουμε πρώτα να αποχωρήσουν όσοι δεν έχουν εργασία.